Λοιπόν, ξαναρχίζουμε και δημοσία και σε ολομέλεια. Ήρθατε όλοι για την, για την ακρόαση σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, παρουσία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Ρούτζι, που είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά. Μα τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σα, κ. Ρούτζι, που την είχαμε ζητήσει, όπω ξέρετε, πολλέ φορέ και με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε εδώ. Εντάχει, να ζητήσω από τους συναδέλφους να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 30ης Μαρτίου. Έχετε παρατηρήσεις? Όχι. Ανακοινώσεις. να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το έργο που έγινε στο Περού. Μετά το 2000 υποστηρίξαμε την δημοκρατική ανάκαψη των χωρών. Μετά από δίκη ο πρόεδρος Φουχημόρη καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Σε πολλές περιπτώσεις του Κοινοβούλιο είχαμε ζητήσει με τα ψηφίσματά μας να ε, αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτά που έγιναν και τη διάρκεια τη προεδρίας του. Για την σύνταξη στη Γάζα, όπως ξέρετε το Συμβούλιο των Δικαιωμάτων Ανθρώπου στη Γενέβη διεύρυνε, και αυτό μας χαροποιεί, το πεδίο εφαρμογής της ε, διεθνούς έρευνας που διεξάγει, όπως ζητήσαμε, έρευνα και ανεξάρτητη και αμερόληπτη για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των ε, επιχειρήσεων ανάμεσα στο Δεκέμβριο του 8 και τον Ιανουάριο του 9 στη Γάζα από όλε τι πλευρέ. Ένα πολύ ε, έντιμο άνθρωπο, ο κ. Ρίτσαρντ Γκόλστον που ήταν πρόεδρο του ε, Διεθνού Δικαστηρίου για την Ρουάντα και την πρώην Ιουγκοσλαβία που ανέλαβε την ε, αποστολή αυτή. Λευκοδοσία. Σα το λέω γιατί είχαμε εξετάσει το ενδεχόμενο να στείλουμε ένα μέλος τη υποεπιτροπή μας στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στη χώρα αυτή. Μετά από κοινή συμφωνία του Προέδρου της Αντιπροσωπείας και του Προέδρου της Επιτροπής Αφέτα κυρώθηκε η επίσκεψη αυτή γιατί με βάση τις προκαταρκτικές συζητήσεις είχε θεωρηθεί ότι δεν ήταν ικανοποιητικέ οι προποθέσει και το επίπεδο των πολιτικών συναντήσεων δεν ήταν αποδεκτό για το Κοινοβούλιο και επιπλέον είχε ζητηθεί να αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών που εμείς είχαμε θεωρήσει ανεπαρκώς ε, διάφανες. Ενώ είχαμε κατακρίνει και την απαράδεκτη στο παρελθόν εκλογική διαδικασία. Αυτές οι δύο απαιτήσει οδήγησαν στην ακύρωση της επίσκεψης και άρα και της δικής μας συμμετοχής. Τουρκμενιστάν. Είδατε ότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει να μην είναι ικανοποιημένο από τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου για το σεμβασμό των έξι κριτηρίων που έχουμε ε, υπερψηφίσει σε πολλές περιπτώσεις και στην Επιτροπή διεθνού Εμπορίου και την έκθεση για την Κεντρική Ασία του κυρίου Οσδεμίδου. Οπότε δεν δώσαμε τη σύμφωνη γνώμη μας για την συμφωνία αυτή ακόμα τώρα. Διάσκεψη του Ντάρμπαν την επόμενη εβδομάδα θα γίνει οι συζητήσεις πριν την διάσκεψη συνεχίζονται ζωηρά. Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την καθοδήγηση του Βελγίου που είναι η υπεύθυνη χώρα για την διεξαγωγή των εργασιών πηγαίνουν προς τα εκεί που θέλαμε την συμμετοχή των κρατών της Ένωσης στη διαδικασία αυτή με μια σαφή βάση που χωρίς να ξανανοίξει το κουτί της Πανδώρας περιλαμβάνει την αυστηρή αξιολόγηση του προγράμματος δράσης που είχε αποφασιστεί στο Τούρμπαν 1. Παρά τις συζητήσεις, ένα πρόγραμμα δράσης ε, για τη μάχη κατά του ρατσισμού και της ε, ε είχε ξεκινήσει και αυτό είναι δουλειά της Ένωσης και του Βελγίου ως επικεφαλής ομάδας της Ένωσης να παραμείνει πρωτοπόρος στην αξιολόγηση του σχεδίου δράσης. Λοιπόν, δημόσια ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον καθηγητή Τζον Ρουτζή, δικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, υπεύθυνου για το θέμα αυτό, τον καθηγητή Γιάνν Βάουτερς, που θα ετοιμάσει μια μελέτη και την οποία θα μας παρουσιάσει σε λίγο μετά από έτοιμά μας για το ίδιο θέμα. Τον κύριο Τζον Μόρισον, παρόντα εδώ, Διευθυντή του Ινστιτούτου Δικαιωμάτων Ανθρώπου στον κόσμο των επιχειρήσεων, την κυρία Ρουθ Καζάλ, συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Δικαιοσύνη στις Επιχειρήσεις και ο κύριος Τζον Evans, όλοι εδώ, εξαιρετικό αυτό. Ο κύριος Τζον Evans είναι Γενικός Γραμματέας Συμβουλευτικού Χαρακτήρα στην Συμβουλευτική Επιτροπή στον ΩΣΑ. Θα ζητήσω από τον κύριο Χάουιτ να έρθει και να παρουσιάσει μια κοινή στα βασικά στοιχεία που πλαισιώνουν την συζήτηση για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Αφού υπενθυμίσω ότι δεν είναι μικρό πράγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε γύρω στις 80.000 επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. αν δεν προσθέσουμε και τις θηγατρικές, που είναι άλλες τόσες, διπλασιάζουμε τον αριθμό. Γύρω στις 80.000 επιχειρήσεις θηγατρικές ευρωπαϊκών δουλεύουν στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για μία από τις βασικές λοιπόν προτεραιότητες του Κοινοβουλίου μας. Κύριε Χάουιτ, έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ δεν θα ακούσουν εμένα. Ε, ευχαριστώ για το ότι οργανώσετε αυτή την, επιτρέψτε να οργανωθεί αυτή η ακρόαση. Αυτό ξεκίνησε από τότε και εσείς πρόεδρε και εγώ. Θέλαμε να φροντίσουμε ο καθηγητής Ράγκη να μιλήσει στο κοινοβούλιο σε αυτή εδώ τη θητεία λόγω της σημασίας που αποδίδουμε στο, στις επιχειρήσεις και το σεβασμό εκ μέρους των επιχειρήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστηρίξαμε την εντολή του Τζον και εγώ προσωπικά συνεργάστηκα προκειμένου να επηρεάσουμε την αντιπροσωπεία μας στην Γενέβη για την εντολή αυτή και με τους νορβηγούς συναδέλφους είναι υπεύθυνοι για την ε, εποπτεία όσον αφορά την επέκταση της εντολής πέρυσι. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να θέλουμε να υπάρξει ένα βήμα για τον Τζον στο Κοινοβούλιο τώρα που τελειώνει η θητεία του και όπως συμφωνήθηκε πέρυσι στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το θέμα επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα έχει σημειωθεί πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικά βήματα έχουν σημειωθεί. Σημαντικό για την ακρόαση είναι πρώτον να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, να γίνει γνωστή η έκθεση αυτή, αλλά επίση και να δούμε τι επιπλέον μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε τι διάφορες συστάσει Έχουμε την ψυχική προεδρία σήμερα και ευχαριστώ για την παρουσία της. Έχουμε εκπροσώπους από την επόμενη τη Σουηδική Προεδρία και ελπίζω ότι φέτος θα είμαστε σε θέση να κινηθούμε από τη θέση όπου τα κράτη-μέλη ψήφισαν και υποστήριξαν στην Γενέβη την έκθεση του Τζον και την εντολή για τον Τζον να περάσουμε στις συστάσεις, στις προκλήσεις που μας τις έχει θέσει επιτάπητος να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι και ουσιαστικά το αντικείμενο της σημερινής ακρόασης. Βέβαια, συζητιέται το θέμα στην Ένωση τι σημαίνει η ευθύνη των επιχειρήσεων. Ίσως δεν είναι ακριβώς το ίδιο επιχειρήσει και ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, κατά κάποιο βαθμό, η συζήτηση ε, και έχουν πολλούς παρόντες εκ μέρους της Κομισιόν η συζήτηση που γίνεται στα όργανα της Ένωσης για την ευθύνη των επιχειρήσεων σωστά να καλύπτει και τη δουλειά που γίνεται από την πλευρά των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Συμβουλίου και του καθηγητή Ράγκη. Αλλά δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και εμείς ως Ένωση και ως κρατημέλη έχουμε υποχρεώσει ως κυβερνήσεις να προστατεύουμε όσον αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα τους εργαζόμενους για επιχειρήσεις που δουλεύουν μέσα στα σύνορά μας. Από την Γενική Διεύθυνση της Εσωτερικής Αγοράς για όλες τις διευθύνσεις για τις ε, εξωτερικές σχέσεις όλοι έχουμε ευθύνες και πρέπει να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις. Έχουμε λοιπόν μια φορτωμένη ημερήσια διάταξη για σήμερα και είμαι περήφανος για το ότι ο Τζον ε, δέχτηκε να έρθει σήμερα να μας μιλήσει. Θα σε ακούσουμε με πάρα πάρα πολύ προσοχή και ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριε Ρούτζη, ήρθε η ώρα σας, η σειρά σας. Πέρυσι κατεφέστε μια έκθεση η οποία υπέστη και κριτική και δέχτηκε και επένους. Αναφερθήκατε στις διάφορε προκλήσει στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και το σεβασμό εκ μέρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτοχρόνω δεν προτείνατε ένα δεσμευτικό νομικό πλαίσιο Αυτά ήταν οι, οι κριτικοί στην έκθεση σα. Σήμερα ετοιμάζεται την επόμενη έκθεση για το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν εύλογο για μας να θέλουμε να ακούσουμε από εσά τον ίδιο εξηγήσει και μετά να συζητήσουμε. Έχετε το λόγο. thank you very much, Madam. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ρίτσαρτ και ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να μετέχω στην ακρόαση αυτή ως πολιτικός επιστήμονας που εξετάζει την εξέλιξη των θεσμών διακυβέρνησης πάντα χαίρομαι που επισκέφτομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση και διδάσκομαι από τις εμπειρίες και τα πειράματα που εφαρμόζεται. Εδώ με φέρατε ωστόσο όχι για να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να μοιραστώ μαζί σας τα αποτελέσματα της εντολής που ανέθεσα που μου ανέφεσαν το 2005 μετά από την, το αίτημα τη τότε επιτροπή Δικαιωμάτων Ανθρώπου στον τότε Γενικό Γραμματέα κύριο Κόφη που όρισε έναν ειδικό αντιπρόσωπο για τι επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζοντα την αυξανόμενη σημασία του ζητήματο. Αυτό που θέλω λοιπόν να κάνω σήμερα είναι να σα ενημερώσω για το πώς έχει τώρα η εντολή και να εξηγήσω σε λίγα λεπτά το αδιέξοδο που αντιμετώπισα και που αντιμετώπισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν το αντιμετωπίσουμε, ίσως να μπορέσουμε, μαζί ίσως να μπορέσουμε και να το λύσουμε. Όπως αναφέρθηκε τον περασμένο Ιούνιο, το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον ΟΗΕ ομόφωνα καλωσόρισε ένα πλαίσιο πολιτικής για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα που είχα υποβάλει. Πρόκειται για συνήθιστη πράξη από δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν ομόφωνη η αποδοχή, κάτι ασυνήθιστο στο, σε μια συζήτηση στο Συμβούλιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεύτερον, για πρώτη φορά ο μηχανισμός του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή και το Συμβούλιο και η Επιτροπή νωρίτερα, έλαβε ουσιαστική πολιτική θέση για τη σχέση επιχειρήσεων και δικαιωμάτων ανθρώπου. Είπε ότι εμεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρούμε ότι τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτική που λειτουργεί και οριοθετεί την συνολική πρακτική και το συνολικό πλαίσιο που θα ακολουθείτε όσο προχωρούμε. Στο ίδιο ψήφισμα το Συμβούλιο, με δεδομένο ότι τίποτα το καλό δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο, παρέτεινε για τρία ακόμα χρόνια τη θητεία μου και μου ζήτησε να κάνω πιο ορθολογικό το πλαίσιο. Τι εννοούσε, να δώσω συγκεκριμένη καθοδήγηση σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα, ιδιαίτερα τα κράτη, τις επιχειρήσεις αλλά και άλλους. Και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε μετά την έγκριση του σχετικού ψηφίσματος. Πρόσφατα έστειλα μια έκθεση προόδου στη Γενέβη με ενημέρωση για το πρώτο έτος σχετικά με το πώς ε, προχωρήσαμε έκτοτε. Θα σας δώσω τώρα εν ολίγης το πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά του πλαισίου αυτού. Διότι οι πληροφορίες από το Συμβούλιο δεν ταξιδεύουν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε χωρίς να βοηθηθούν λίγο. Το πλαίσιο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος, η υποχρέωση του κράτους. Υποχρέωση. Και λέω υποχρέωση εσκεμένα γιατί υπάρχει και νομική υποχρέωση εν μέρει. Η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι τρίτοι. Μεταξύ αυτών είναι και οι επιχειρήσεις. Όταν ένα κράτος υιοθετεί εργαλεία δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, υιοθετούν και μία υποχρέωση να προστατεύουν την, από την παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο όταν αυτή η παράβαση διαπράττεται από τα κράτη αλλά και από άλλες πλευρές π.χ. τις επιχειρήσεις που μπορεί να, να παραβιάσουν τα δικαιώματα αυτά. Αυτό είναι νομική υποχρέωση βάσει της διεθνούς, ε, του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν πολύ, πολλές επιπλοκές. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η εξοεδαφική ε, δυνατότητα ε, καταστολής και τιμωρία των παραβιάσεων αυτών. Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει αυτή η εξοεδαφική αρμόδια των κρατών. Είναι ένα πρώτο ζήτημα. Δεύτερο θέμα. Η ευθύνη των επιχειρήσεων να σεβαστούν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτό το λέμε ευθύνη και όχι καθήκον, διότι δεν υπάρχει διεθνής νομοθεσία που να εφαρμόζεται ευθέως στις επιχειρήσεις πέραν κάποιων πολύ στενά οριζόμενων τομέων όπως ε, τα διεθνή, η διεθνής εγκληματικότητα. Ωστόσο, άποψή μας είναι ότι οποιαδήποτε εθελοντική πρωτοβουλία που γνωρίζουμε, είτε το Παγκόσμιο Σύμφωνο, είτε είναι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων, είτε είναι δηλώσει του διεθνού Εμπορικού Επιμετηλίου, είναι δηλώσει του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασίας, είναι δηλώσει του ΟΣΑ, όλα τα κείμενα αυτά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Λένε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει ή οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και να σέβονται σημαίνει στην ορολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην επεμβαίνουν, να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων καθώς ασκείς τις δραστηριότητές σου. Η προσέγγιση μας λοιπόν προς αυτό το θέμα ήταν να δεχθούμε αυτά που μας λέει η επιχειρηματική κοινότητα. Για ότι σέβονται δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο τους ρωτάμε πώς το ξέρετε αυτό. Πώς ξέρετε ότι σέβεστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως επιχείρηση, ως όμιλος, έχετε κάποιες δομές, κάποιο πλαίσιο που θα σας επιτρέψουν να αποδείξετε και στους εαυτούς σας και στους εξωτερικούς ελεγκτές ότι σέβεστε όντως τα ανθρώπινα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρευνες των πράξεων των επιχειρήσεων δείχνουν και αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες επιχειρήσεις τέτοια συστήματα δεν υπάρχουν. Άρα, στην έκθεση που αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, πέρυσι, που θέσαμε τα βασικά στοιχεία αυτού που αποκαλούμε η υποχρέωση των ε, επιχειρήσεων να τηρούν την δέουσα επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα. Το, το τρίτο θέμα είναι η πρόσβαση στην νομική θεραπεία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα είχαν νόημα αν δεν υπήρχε πρόσβαση σε ε, ένομη προστασία για τα θύματα. Τα, η καλύτερη ενημέρωση των κρατών και των επιχειρήσεων στην εργατική νομοθεσία είναι τα συνδικάτα, αλλά σε ό,τι αφορά τις τοπικές κοινότητες ή τις αυτόνομες κοινότητες, οι μηχανισμοί ενημέρωσης των ε, ε, κατοίκων αυτών δεν προχωρούν γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση, ε, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει δομή στις επιχειρήσεις που να δέχεται κάτι τέτοιο ενώ ταυτόχρονα η δικαστική προστασία είναι ανύπαρκτη τελείως περιορισμένη. Τρεις βασικές αρχές. Υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από την κατάχρηση από τρίτους με και, και των επιχειρήσεων βέσεων και νομοθετικά και ρυθμιστικά. Δεύτερον, ευθύνη των επιχειρήσεων να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατά βάση σημαίνει να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων και να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο με την εφαρμογή της δέωσης επιμέλειας στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρίτον η ενίσχυση των μηχανισμών ε, θεραπείας είτε δικαστικής είτε εξωδικαστικής σαν τμήμα και της υποχρέωσης του κράτους να προστατεύει και της ε, ευθύνη των επιχειρήσεων να μην παραβιάζουν. Αυτές οι τρεις, αυτοί οι τρεις πυλώνες λειτουργούν συντονισμένα, όχι απομονωμένα. Επίσης, καθιστούν σαφές ότι οι υποχρεώσεις των κρατών διαφέρουν ουσιαστικά από την, τις ευθύνες των επιχειρήσεων. Στο παρελθόν, πολλές, ευ, πολλές προσπάθειες όπως οι κανόνες για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν μπερδέψει ή είχαν αναμίξει τις υποχρεώσεις των κρατών και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε τέτοιο βαθμό που δεν ήταν δυνατόν να πούμε ποιος ήταν υπεύθυνο γιατί στην πράξη. Και εν τέλει, θα να Το μόνο που υπήρχε συμφωνία ήταν να κατηγορεί ένα τον άλλον. Όχι η δική σου δουλειά είναι, όχι η δική σου δουλειά είναι. Τώρα προφανώ υπάρχει μια διαφοροποιημένη ευθύνη και υποχρέωση των κρατών και διαφορετική των επιχειρήσεων. Συμπληρωματικέ ωστόσο. Αυτές είναι οι αρχές. Τώρα πώς παρουσιάζουμε τα συστατικά τους. Λίγα παραδείγματα θα δώσω πρόεδρε, δεν θέλω να παρατείνω γιατί καλό θα είναι να κάνουμε μια συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Η υποχρέωση του κράτους να, παρέχει προστασία. Οι επιχειρήσεις ξέρανε εδώ και πολλά χρόνια ποιες ήταν ε, οι υποχρεώσεις στον τομέα της κατάχρησης των δικαιωμάτων ανθρώπου στον τομέα των σχέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρήσεων το πράγμα ήταν ωστόσο λίγο πιο ασαφή. Οι περισσότερες χώρες σε κάποιους βασικούς τομείς όπως εργασιακέ προδιαγραφές, απαγόρευση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας έχουν θεσπίσει πολιτικές, κανονισμούς και θεσμικά όργανα. Ξέρουν πάνω κάτω τι αναμένεται από αυτούς. Ε, το Παγκόσμιο Γραφείο Εργασία Φρύμπιν βοηθάει σημαντικά. Πέραν αυτών των βασικών τομέων, αυτό που βρήκαμε στην έρευνα μεταξύ κυβερνήσεων είναι αυτό που αποκαλούμε η πολιτική, οι ασυνέπειες πολιτικών. Σε δύο κατηγορίες. Κάθετες ασυνέπειες. Μία χώρα προσχωρεί σε ένα νομικό εργαλείο δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς να ξέρει ή να ενδιαφέρεται τις συνέπειες που έχει η προσχώρησή της αυτή στην εφαρμογή του κειμένου, το οποίο ποτέ δεν ε, εφαρμόζεται. Και αυτό τον, ε, αυτή τη συμπρακτική την ονοματίζουμε με ευγενικό τρόπο κάθετη ασυνέπεια. Υπάρχει ωστόσο και οριζόντια ασυνέπεια που εμφανίζεται και σε πολλές προοδευτικές λεγόμενες χώρες. Δηλαδή, προσπαθούν να δώσουν μια πολύ στενή οριοθέτηση του όρου επιχείρηση και ανθρώπινα δικαιώματα που είναι με ένα γραφείο, ένα μικρό γραφείο στη, στον κυβερνητικό μηχανισμό. Υπάρχει μια μονάδα η οποία ασχολείται με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν ωστόσο μια χώρα νομοθετεί ή όταν ε, η κυβέρνηση ασχολείται με θέματα ε, διακυβέρνηση επενδυτικών ε, νομοθεσιών κλπ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα χάνονται, δεν υπάρχουν. Οι δεσμεύσει λοιπόν που αναλαμβάνει ένα κράτο να προστατεύσει από την παραβίαση των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν περνάνε ποτέ σε πολιτικές και σε νομικά κείμενα που επηρεάζουν ευθέως τις επιχειρήσεις. Ε, εταιρικό δίκαιο, εμπορικές συμφωνίες, επενδυτική νομοθεσία, επενδυτικές συμφωνίες, όλα αυτά δεν έχουν μνήα για ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μικρή οριζόντια εισχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις πολιτικές. Ο κύριος στόχος μας λοιπόν στην εντολή που θέλουμε να προχωρήσουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα αλλάξει. Συνεργαστήκαμε λοιπόν στενά με ένα δίκτυο δικηγόρων που ασχολούνται με, εταιρικέ, με εταιρικό, εμπορικό δίκαιο και καλύπτουν τέσσερις διαφορετικές ε, ένομες τάξεις ζητώντας να δούμε πώς αυτή τη στιγμή ε, η εταιρική νομοθεσία τα δικαιώματα των διευθυντών, των διευθυντών μπορούν να επέμβουν ή να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν την κυβερνητική πράξη. Επίσης εξετάσαμε μια σειρά ε, διμερών εμπορικών επενδυτικών συμφωνιών ή διακρατικών συμφωνιών για να δούμε πώς μπορούν να περιορίσουν τη δυνατότητα επέμβαση των κρατών γιατί με βάση τις συμφωνίες αυτές μια επιχείρηση ε, μπορεί να καταγγείλει το κράτος εάν θεωρεί ότι μια νομοθεσία καινούργια επηρεάζει την κερδοφορία της. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, η κυβέρνηση της Αφρικής βρίσκεται σε διεθνή διαιτησία ε, όπου την παρέπεψε μια εξωτερική ιταλική βιομηχανία που θέλει να αποζημιωθεί για τις οικονομικές συνέπειες της νομοθεσίας για την ε, πολιτική ανάδειξη της ε, πλειοψηφίας των μαύρων, το Black Empowerment Act. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Αν η Νότιο Αφρική μετά την ε, περίοδο του Παρχάη δεν μπορεί να υιοθετήσει νομοθετικά κείμενα για να προωθήσει τα δικαιώματα τη πλειοψηφία ε, του, πληθυσμού Χωρί να φοβάται ότι θα αποζημιώσει με σημαντικά ποσά ε, μια Ιταλική εταιρεία, κάπω πρέπει να αλλάξουν οι συμφωνίε επενδύσεων. Και το βλέπουμε αυτό προσπαθώντας να παράσχουμε κάποιες βασικές καθηγητήριες γραμμές στην διαμόρφωση των επενδυτικών ε, συμφωνιών. Ένα τρίτο παράδειγμα. Υποχρέωση προστασία εξωτερικού του κράτους. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το καθεστώ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω έχει είναι δυνατόν να λειτουργήσει με την πρόθεση που προβλεπόταν σε ζώνες όπου υπάρχει μια σύραξη, όπου υπάρχει ένας φίλος πόλεμος, Ωστόσο, στέλνουμε επιχειρήσεις στις χώρες αυτές και προωθούμε επενδύσεις για καλό σκοπό, γιατί μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά οι αξιολογικές εταιρείε για τις εξαγωγές και αυτοί που προωθούν επενδύσεις, προωθούν επενδύσεις στις περιοχές αυτές χωρίς να ζητάνε την αυξημένη αυτή πρόνοια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου και ωστόσο ένα ίδρυμα το οποίο αξιολογεί μια επένδυση δεν απαιτεί κάτι παραπάνω από ότι αν παραδείγματος χάρη κάποιος θα επένδυση δανεία. Δεν χρειάζονται επιχειρήματα για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι νομικό θέμα ή είναι κάτι άλλο. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά, για μην πω τίποτα βαρύτερο. Χρησιμοποιούνται κυβερνητικά κονδύλια για να αυξηθεί ο κίνδυνος κατάχρησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτά ήταν μερικά παραδείγματα που τα κοιτάμε κάτω από την τίτλο αυτό «Υποχρέωση του κράτους». Τώρα το δεύτερο για την ευθύνη σεβασμού, responsibility. Ποιες είναι οι συνιστώσεις αυτής της ε, δέουσας προσοχής, due diligence, πώς εφαρμόζεται στις διάφορες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, για τράπεζες που δανείζουν αλλά δεν λειτουργούν οι σε ένα πρόγραμμα. Σχετικά δηλαδή με την εφαρμοσιμότητα των γενικών αρχών της ε, ε, οφειλόμενης προσοχής, due diligence. Αυτά πάντα για το δεύτερο πυλώνα. Και έρχομαι στον τρίτο πυλώνα τώρα πάλι, στην αποκατάσταση, στη διόρθωση, στη θεραπεία. Rehabilitation. Στο δικαστικό σκέλος, που είναι και το πιο δύσκολο και θα επανέλθω σε αυτό, αυτό που κάνουμε είναι κοιτάμε ποια είναι τα εμπόδια. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις. Ξέρουμε ποια είναι τα εμπόδια πρόσβαση στη δικαιοσύνη στις περισσότερες χώρες του. Ξέρουμε. Τα περισσότερα από αυτά φυσικά είναι και εμπόδια και για τα θύματα κατάχρησης εκ μέρους των επιχειρήσεων. Όμως, ειδικά για τις επιχειρήσεις υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Πάμε χάρη όσον αφορά την ε, υπερεθνική συνεργασία λόγω της διαφορετικού νομικού προσώπου, νομικής προσωπικότητας. Τις ιδιότητες του, του προσώπου ως προς την επιχείρηση. Επίσης, έχουμε και την, ε, το μη δικαστηριακό χώρο. Γιατί εκεί είναι δυνατόν να έχουμε πιο γρήγορη πρόοδο. Και αυτό μετράει πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη συνεργαζόμαστε με τις ενώσεις, ε, διεθνείς ενώσεις υποχρεώσεων και επιμέρους υποχρεώσεις για πιλωτικά προγράμματα, για μηχανισμούς καταγγελίας παραπώνων ως προς την επιχείρηση. Εμείς δίνουμε τα κριτήρια, τις παραμέτρους, τις αρχές με βάση τις οποίες θα λειτουργεί το σύστημα, το υποπτεύουμε το σύστημα και οι κοινότητες που πλήττονται από δραστηριότητα μιας επιχείρησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό, το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό, ε, για να καταγγείλουν και για να διδαχθούν. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι ο κόσμος συνήθως δεν ξέρει πού να πάει όταν έχει ένα παράπονο, μια καταγγελία. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα γουίκι, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες της επίσημης κοινότητας και μπορεί να βοηθεί ένα, ένα άτομο που είναι θύμα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις με μια μορφή αλληλοδραστική online σε σχέση με καταγγελίες έναντι επιχειρήσεων. Μπορεί να δει κανείς οι κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ. Τι έχει γίνει ως τώρα. Ποιος θεσμός για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τι επιτυχίες έχει, αν έχει ένα τέτοιο είδο πρόβλημα, σε ποιο να κλπ. κλπ. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο. Στην εξοδικαστηριακή διαδικασία. Αυτά κύριε Πρόεδρε με πολύ αδρές πινελιές για το πλαίσιο αυτά που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι στρατηγικές αποφάσεις, κατευθύνσεις που χαράκτηκαν. Όπως είπα και στην αρχή, πριν κλείσω την εισαγωγή μου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που επηρέασε τη συζήτηση και στην Ένωση και όσον αφορά την εντολή που είχε ανατεθεί σε μένα σχετικά με την διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών μέτρων. Νομίζω την έχετε ακούσει αυτή τη συζήτηση. Πώς γίνεται στην Ένωση. Κατ' εμέ, η ίδια η συζήτηση είναι τόσο στήρα, θα έλεγα και μη παραγωγική, που δεν αξίζει να συζητάμε πια. Ωστόσο, υπάρχει μία συνιστόσα που δεν συζητήθηκε αρκετά και που αποτελεί εμπόδιο στην δημιουργική σκέψη και δράση. Όλοι συμφωνούμε ένα μείγμα προαιρετικών και υποχρεωτικών μέτρων είναι κάτι που απαιτείται. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις και άλλα συναφή όργανα και οργανισμοί συνήθως δεν εκτιμούν απόλυτα το ρόλο τους ακόμα και όταν προωθούν προαιρετικές λύσεις. Μερικές κυβερνήσεις και οργανισμοί λένε αποφασίσαμε ότι αυτό θα είναι προαιρετικό, τέλειωσε η δουλειά μας. Αυτό είναι σόφισμα. Δημιουργεί προβλήματα. Πρακτικά. Θα σας αναφέρω τρία σενάρια για να καταλάβετε γιατί μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Πρώτο, Δεν γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ στόχων πολιτικής από τη μια και των μέσων υλοποίησης αυτής της πολιτικής και των στόχων. Ας υποθέσουμε έναν ευρύ ορισμό της Ένωσης του CSR. Είναι μια έννοια με βάση την οποία με επιχείρηση ενσωματώνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις δραστηριότητές της και στην σχέση της με τους μετόχους της σε προαιρετική βάση. Ωραία. Αυτός είναι ο ορισμός. Ας υποθέσουμε ότι μία υποθετική μονάδα ε, αποφασίζει να δράσει με βάση αυτόν τον ορισμό ενώ κρατική, κρατικός οργανισμός. Ο στόχος είναι οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν αυτά τα κριτήρια κοινωνικά και περιβαλλοντικά που να αντικατοπτρίζουν υποτίθεται την ανάγκη της εταιρεία να σέβεται οι κοινωνικές ε, ε, προδιαγραφές και κανόνες και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός είναι ο στόχος. Το μέσον, το προτιμόμενο μέσον είναι προαιρετικό. Άλλο στόχος, αλλά το μέσον. Βέβαια αυτοί που επικρίνουν τις προαιρετικές δράσεις θα πούνε με αυτά τα μέσα δεν μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο. Αυτό δεν το συζητάω. Υποθέτω τι γίνεται. Παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το εξή. Επαφίεται σε κάθε εταιρεία να αποφασίσει μόνη της ποια κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και μελήματα είναι τα πιο σημαντικά και τι σημαίνει τα ενσωματώνω. Αν δεν τους δοθεί περιττέρω καθοδήγηση στις εταιρείες Παίρνουν λοιπόν οι επιχειρήσεις χωρίς καθοδήγηση αποφάσεις. Ο στόχος αρχίζει και αυτός να μπαίνει λίγο στα προαιρετικά χωράφια. Γιατί κάθε επιχείρηση αποφασίζει μόνη της τι σημαίνει αυτός ο όρος, τι σημαίνουν αυτά τα κριτήρια, τα μελήματα. Και τι καλούνται να κάνουν οι επιχειρήσεις. Τελικά λοιπόν έχουμε ένα προαιρετισμό 100% και στα μέσα αλλά και μέσω της αυτοερμηνίας και του στόχου. Αποτέλεσμα δεν έχει πολιτική. προσδοκίες άλλων κοινωνικών εταίρων. Άρα έχουμε λοιπόν με προαιρετική πολιτική CSR τι θα υπάρχει εκεί μέσα. Ποιες είναι οι προθέσεις αυτής της πολιτικής. Τι ελπίζουμε να πετύχουμε. Να νιώσουμε κοινή κατανόηση για τους έννοιες κλειδιά. Τι σημαίνει ενσωματώνω. Είναι μια δημόσια λειτουργία να εξηγήσουμε τι σημαίνουν αυτά. θα έπρεπε να απαιτεί η υποστήριξη μιας διαδικασίας ε, χθενίσματος κατά κάποιο τρόπο κοινωνικού που θα ορίζει ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Δεν αρκεί να πούμε αφήνουμε ποιες είναι οι, βελτιές, οι βέλτιστες πρακτικές. Αυτό είναι μια κοινωνική κριτική και οι δημόσιες αρχές πρέπει να ασκούν αυτή τη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο, αλλά όλες οι πολιτικές CSR δεν πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια του να αποτελούν πολιτική με αυτή την έννοια. Επειδή υπάρχει ο φόβος να μην τυχόν κινηθούμε πέραν του προαιρετικού. Δηλαδή τι θέλω να πω. Μία αντίληψη του τι σημαίνει υποχρεωτικό και τι σημαίνει προαιρετικό και ένας περιορισμένος ορισμός τι σημαίνει προαιρετικό μπορεί να μας πάει πέραν του προαιρετικού αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση, προς το laissez-faire κατεύθυνση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία ας πούμε δέκα χρόνια στην Ένωση. Δεύτερο σενάριο. Φόβος μην τυχόν πάμε πέρα του στενά ορισμού του προαιρετικού χώρου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τη δημόσια αρχή στο να αυξήσει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Δεν την εξυπηρετεί την επιχείρηση αυτό. Πάμε χάρη. Ζώνε όπου υπάρχει σύραξη στρατιωτική. Μια επιχείρηση θα ήθελε να έχει μια κατεύθυνση από την χώρα την οποία προέρχεται από μια διεθνή, διεθνή οργανισμό να, πώς να αποφύγει να εμπλακεί μέσα στη σύρεξη αυτή ή να γίνει ε, συνεργός σε κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πάρα πολύ κοινό σε περιοχές που σοβεί τέτοιου είδους στρατιωτική δράση. Ο ΩΣΑ έχει ένα εργαλείο αξιολόγησης των κινδύνων, αλλά συνήθως αυτό που χρειάζεται επιχειρήσεις ε, είναι πληροφορίες σε χρόνο μηδέν που μπορεί να δώσουν οι πρεσβείες. Ποια ποια στρατιωτική παράταξη κάνει τι, πού βρίσκεται και πώς μπορεί να αποφύγει η επιχείρηση των κίνδυνο να εμπλακεί στα τεκτενόμενα. Συνήθως οι κυβερνήσεις δεν δίνουν τέτοιο είδους υποστήριξη. Θέλουν να προωθήσουν τις επενδύσεις, άσχετα του, αν, του τι και τι αν υπάρχουν κίνδυνοι. Και το τρίτο σενάριο, ένα πραγματικό δίλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Όταν λειτουργούν σε χώρες όπου η εθνική νομοθεσία έρχεται σε σημαντική αντίφαση, δίνει μικρότερη προστασία από ό,τι διεθνείς κανόνες. Ο Τζον το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει τις επιχειρήσεις και αλλού για την ισότητα των φύλων, για την ε, ελευθεροτυπία και την ελεύθερη έκφραση στο ίντερνετ και στις τηλεπικοινωνίες. Μια χώρα θέλει να λογοκρίνει μια επιχείρηση η οποία είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης πληροφορία. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή. Τι περιμένουμε από μια επιχείρηση σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, οι επιμέρους επιχειρήσεις φυσικά μόνε του δεν μπορούν να το λύσουν αυτό το δίλημα, πρόβλημα. Δεν γίνεται, δεν μπορούν. Χρειάζεται συλλογική δράση. Αλλά η συλλογική δράση των επιχειρήσεων και αυτό είναι πρόβλημα. Οι εταιρείε που δουλεύουν στο Ιντερνετ έχουν ρίξει τώρα μια σειρά από αρχέ. Χρειάστηκε χρόνο, αλλά πολύ λίγε επιχείρησει έχουν υπογράψει αυτόν τον κατάλογο. Περιμένουν βοήθεια από τη μητρικό κράτο. Αλλά το μητρικό κράτο κρατά τα χέρια του μακρά είναι ραδιενεργό υλικό και αφήνει τι εταιρείε μόνε του στα γκάθια να δώσουν τη μάχη αυτή επειδή φοβόνται. Αλλά είναι αυτό είναι προαιρετικό. Πολύ περισσότερα πράγματα μπορεί να γίνουμε στον χώρο του προαιρετικού χωρίς να παραβιαστεί η δέσμευση που έχουμε έναντι του προαιρετικού. Αν επιχειρήσεις ήταν βοήθεια. Είναι ασφαλές νομίζω να θεωρήσουμε ότι αυτό παραμένει στο χώρο του προαιρετικού. Και τελειώνω με δύο σχόλια. Η διεθνής κοινότητα. Είμαστε ακόμα στην αρχή προκειμένου να εγκροθεί το καθεστώς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το καθολικό, το οικουμενικό, για προστασία και ατόμων και κοινοτήτων έναντι καταχρήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από επιχειρήσεις. Ένα είναι σαφές ήδη από τώρα όμως. Το business as usual, δηλαδή μην κάνουμε τίποτα, δεν βοηθάει κανέναν, ούτε καν τις επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην γίνεται τίποτα. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και σύντομα θα τρακάρουμε σε τείχο. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Αυτό σημαίνει να εγκαταλείψουμε ε, ε, στήρες αντιλήψεις που σημαίνουν προαιρετικά ή υποχρεωτικά μέτρα και να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει η συνέργεια των μέτρων και των μέσων. Και δεύτερο, το πλαίσιο θεραπείας που έχει ψηφίσει το Συμβούλιο Εθνικών Δικαιωμάτων δίνει μια πλατφόρμα, μια κοινή πλατφόρμα όπου μπορεί να γίνει μια διαφοροποίηση των συμπληρωματικών υποχρεώσεων και ευθυνών των κρατών ε, ε, ε καθήκοντα των, κυβερνήσεων και ευθύνη των επιχειρήσεων. Κατά από αυτή την ομπρέλα λοιπόν παρέχεται μια έμπνευση κατευθύνσεις και προς κράτη και προς ομάδες κρατών για τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στις συνταγές τις οποίες γράφουν για το τι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, ένα κοινό πλαίσιο είναι. Στο τέλος φυσικά θα έχουμε μια πιο συστημική παρέμβαση από ό,τι έχουμε στο παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν είχαμε μικροκομμάτια λύσεων ασυνάρτητα, ασύνδετα μεταξύ τους σιγά σιγά προχωράμε σε συστημικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καινοτόμο και σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρούτζι. Πρόκειται για μια σαφέστατη και πολύ βούληση αρχική προσέγγιση. Μετά συνεχίζουμε με την παρουσίαση της έκθεσης του κυρίου Βάουτερς. Έχουμε μία ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Παρακαλώ να είσαστε λυτοί, συνθετικοί και αποτελεσματικοί, όπως και είστε κύριε Βόρτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ακολουθήσω τις οδηγίες σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι τιμή σήμερα που είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω βασικά ευρήματα του briefing paper που ετοιμάσαμε για το κοινοβούλιο το οποίο έγινε τελικά 40 σελίδες αλλά δεν είναι και πολύ briefing μάλλον μελέτη στηριζόμαστε στις γενικότερες ε, διεθνείς συζητήσεις κάτι που ήδη μας περιέγραψε πολύ σωστά ο κ. Ράγκη επίσης στη μελέτη αναλύουμε την κατάσταση της πολιτικής των πολιτικών διαργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και την ανάλυση των εξωτερικών διαστάσεων στον τομέα αυτό με υποβολή προτάσεων πολιτικής. Εγώ θα δώσω έμφαση κυρίως στις συστάσεις μας προς την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Το κύριο έβριμα στη μελέτη είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία από, από, από πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προσανατολίζονται στα κράτη και τον ρόλο των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης που είναι το βασικό στοιχείο της πολιτικής για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Στην... Εδώ έχουμε μια σειρά σχολείων και συστάσεων. Όντω η εξωτερική πολιτική τη Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει μέσω του mainstreaming τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις αναπτυξιακές και εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης, στις γενικευμένε προτιμήσεις και στο GSP+, Plus και στην ε, ημερήσια διάταξη του διεθνού Γραφείου εργασία. Ωστόσο, η πρόθεση των δικαιωμάτων ανθρώπου μέσω των εξωτερικών αυτών πολιτικών χρησιμεύει, λειτουργεί μέσω του διαλόγου και των κινήτρων προς τα κράτη που έχουν κακή ιστορία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς λέμε στο σημείο αυτό ότι το θέμα των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν εντάσσεται παρκώς στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Η εξωτερική πολιτική στηρίζεται υπερβολικά στην πολιτική της Ένωσης για την εταιρική ευθύνη που χρησιμοποιείται συχνά σε κείμενα εξωτερικής πολιτικής σαν ένας δρόμος ε, υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δράσεις. Επιπλέον, όπως και ακούσαμε, οι πολιτικές της Ένωσης καταγγέλλονται ως υπερβολικά εθελούσιες, ως ε, στηριζόμενες στην αγορά και ε, στηριζόμενες στις διεργασίες, την ε, την ευθύνη, την λογοδοσία και οι πολιτικές της Ένωσης δεν έχουν υλοποιήσει επαρκώς τις ε, υφιστάμενες πρωτοβουλίες. Οι καταναλωτές δεν μπορεί να καταλαβαίνουν τι σημαίνουν και ποιες, ποια προσθέμενη αξία έχουν. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο να υπάρξει και μια εξορθολόγηση, ούτως ώστε η εταιρική συμπεριφορά να είναι πιο κατανοητή και προσβατή στους κατανοητές και το κοινό. Μετά τα ευρήματα αυτά υποβάλλουμε κάποιες συστάσεις πάνω σε δύο βασικές γραμμές. Πρώτον, ανάληψη συγκεκριμένης δράσης σε διεθνές επίπεδο από την Ένωση και μετά τις συστάσεις της έκθεσης του κ. Ράγκη για το 2008 και των σχετικών συζητήσεων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεύτερον συστάσεις για το κοινοτικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Θα, ας πω πρώτα στο πώς η Ένωση θα μπορούσε να συμβάλλει στην πρόθεση σε διεθνές επίπεδο της ευρωπαϊκής ατζέντα. Έχουμε δύο κυρίες κατηγορίες συστάσεων αφενός συνιστούμε να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε σαφή σε ένα σαφές και διεθνές νομικό πλαίσιο για τις ευθύνες και υποχρεώσεις των εταιριών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο, η δεύτερη κατηγορία συστάσεων εδώ είναι να εθαρρύνουμε την ΕΕ να παραμείνει προπομπός, πρωτοπόρος στις διεθνείς οργανώσεις όσον αφορά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εταιρικά θέματα. Επιτρέψτε μου σύντομα να αναφερθώ σε αυτά, Πρόεδρε. Πρώτον, η ΕΕ υιοθέτησε τη θέση το 2008 στο Συμβούλιο στη Σύνοδο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ότι δεν έβαιναν καλά τα πράγματα σε σχέση με την διεθνή τάξη πραγμάτων από νομικό πλαίσιο. Και εμεί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πιο αναγκαίο αυτή τη στιγμή για τα εταιρικά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ορισμοί σαφών νομικών υποχρεώσεων των εταιριών θα τερμάτιζε εικασίε και οικοτολογίε και αμφίσιμε θέσει και τοποθετήσει από μια ολόκληρη σειρά εμπλεκομένων σε αυτά τα θέματα και επειδή έχουμε και επικρίσεις σε σχέση με την έκθεση του ε, ειδικού απεσταλμένου που αφορά αυτό το θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη ενός σαφούς πλαισίου εταιρικών υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να είναι υποφελές και στις εταιρείες αυτές καθώς και θα μείωνε την αβεβαιότητα την νομική και θα οδηγούσε σε ένα ε, σταθερό πλαίσιο και γι' αυτό θα δίνουμε στην έκθεσή μας πρώτα απ' όλα η ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την εντολή και το στόχο του ειδικού εντεταλμένου, όχι μόνο με κονδύλια, αλλά επίσης ενθαρρύνοντας να επικεντρωθεί περισσότερο και να προσέξει περισσότερο την ανάπτυξη δεσμευτικών διεθνών κανόνων όσον αφορά αυτά τα θέματα, όσον αφορά τον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη αυτή την αλυσίδα, σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερη σύσταση προς την ΕΕ. Η ΕΕ να είναι αρρωγός, είναι στοχεύσει στην ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για την προστασία επενδύσεων πράγμα που πρέπει να οδηγήσει φυσικά στην προστασία επενδυτών, αλλά επίσης να δίνεται η δυνατότητα ώστε η συνιστόσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καλύπτεται και να λαμβάνεται υπόψη. Αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα για να ισορροπήσουμε τα δύο σκέλη, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματο θα πρέπει κανείς να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι η χώρα υποδοχής θα συνεχίσει να έχει ένα δικό της αριθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως εδώ υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, κάνοντας λόγο για αυτό το νομικό πλαίσιο που πρέπει να αναπτυχθεί για την προστασία επενδύσεων. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα εδώ, το θέμα της λογοδοσίας των επενδυτών όσον αφορά τις περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ενδιαφέρον ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει νέες αρμοδιότητες και εξουσίες όσον αφορά το επίπεδο της κοινή εξωτερικής εμπορικής πολιτικής που αυτό σημείο εφεξής για την προστασία των επενδυτών και επενδύσεων θα δίνει ευκαιρία να καλύπτονται όσον ε, αφορά κιόλα και τι αυξημένε αρμοδιότητε τη Ευρωβουλή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα στο μέλλον. Επίση, συνιστούμε η ΕΕ να συνεχίσει να προσπαθεί να αποσαφηνίσει τα πράγματα σε θέματα όπω και την δυνατότητα, για παράδειγμα, να υπάρξει δίωξη, να υπάρξει προσαγωγή στα δικαστήρια τέτοιων εταιριών αν υπάρχουν παραβιάσεις ε, διεθνούς ε, ανθρωπιστικού δικαίου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μπορεί με μια να υπάρχουν πραγματιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά την κοινή προσέγγιση δίωξης εγκλημάτων όμως δεν βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο το σημερινό της δίωξης ή του κώδικα ε, για τα εγκλήματα και νομίζω πρέπει να εμείνουμε και να επιμείνουμε να δοθεί συνέχεια σε αυτό. 11 χρόνια μετά από τις διαπραγματεύσεις του καθεστώτος ε, του δικαστηρίου για, μέσω της, ε, των διαβουλεύσεων της Ρώμης για τη συνθήκη της Ρώμης είναι σημαντικό να δώσουμε συνέχεια. Τέλος είναι σημαντικό επίσης να δώσει μια αποσαφήνιση του καθεστώτος των εργατικών διατάξεων ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά φυσικά το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνοντας συνέχεια στις προσπαθίες της. Επίσης άλλη σύσταση σε διεθνές επίπεδα είναι να ενθαρρύνουμε την ΕΕ να ενθαρρυνθεί να συνεχίσει να να έχει ρόλο προπομπού πρωτοπόρου σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκόσμια και σε εκείνους τους διεθνείς οργανισμούς που δραστήρια συζητούν και διαβουλεύονται για αυτά τα θέματα και από τον κύριο Ρούντι αναφέρθηκε επίσης ότι σε σχέση με τις συζητήσεις για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νομίζουμε ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να πιέσει ώστε να υπάρξουν πιο φιλόδοξα βήματα και μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτά τα επίπεδα. Υπάρχουν όμως και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και φόρα όπου αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, όπου θα μπορούσε η ΕΕ να ξεκινήσει μια διαβούλευση, για παράδειγμα όσον αφορά τον ΟΣΑ, για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών, όπως ε, ε, αναφέρεται επίσης και στην έκθεση του κυρίου Ρούτζι και έτσι με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρει ώστε να αξιολογήσουμε την εξέλιξη, μετεξέλιξη αυτών των πρακτικών σε αυτό το επίπεδο και να επικεντρωθούμε και στο θέμα της λογοδοσίας, της υπευθυνότητας εταιριών όσον αφορά αυτές ε, τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που εκκρεμούν. Με το ε, Διεθνές Γραφείο Εργασίας για παράδειγμα, ακόμα και με τον ΠΟΕ, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπου το θέμα θα μπορούσε να είναι πώς θα μπορούσαν να συγκεραστούν ε, τα θέματα διατάξεων και προδιαγραφών αυτών των ε, οργανώσεων ή οργανισμών όσον αφορά πάντα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την άλλη πλευρά. Έχουμε ένα δεύτερο κεφάλαιο στην έκθεσή μας που περιέχει μια σειρά συστάσεων που αφορούν την ε, χρήση ε, για τις ίδιες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσέγγιση τη νομική όσον αφορά τα θέματα εταιριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν εκεί συστάσεις ε, και ξεκινάμε με μια πρόσκληση να επανεξεταστεί η εθελούσια εφαρμογή ή ε, προσέγγιση όσον αφορά την CSR, την ΕΚΕ, την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και αυτό επειδή φυσικά είναι θέματα σημαντικά αυτά όσον αφορά τα εταιρικά ζητήματα και πρέπει να συμπληρώνονται από μια πιο δεσμευτική προσέγγιση και όχι μόνο εθελοντική και για τα θέματα της λογοδοσίας επίσης ε, των εταιριών όσον αφορά παραβιάσεις ε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι ενθαρρύνουμε και συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει την πολιτική της για την ΕΚΕ, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ώστε να εντοπιστούν και να προσαφινιστούν με σαφέστερο τρόπο υποχρεώσεις για τις εταιρείες και να υπάρξουν τρόποι ώστε να λογοδοτούν οι εταιρείες σε περίπτωση παραβάσεων ή παραβιάσεων. Επίσης αναφέρθηκε πιο πριν η, ΕΚΕ, η εταιρική κοινωνική ευθύνη επικεντρώνεται σε κάποιες διαδικασίες, σε διεργασίες. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα και να μπορούμε να συναγάγουμε τα καλύτερα μαθήματα από αυτά τα συμπεράσματα όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, best practices. Επίσης όσον αφορά την Ευρωβουλή που επανειλημμένα το είχε προτείνει, νομοθεσία να δημιουργηθεί ώστε να υπάρξει υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης και τα θέματα της ε, ε, συνέχειας που, δίνονται, που δίνεται. Και αυτό θα πρέπει σε σχέση με τους κανόνες που θα θεσπιστούν να εξεταστεί και με τους ε, consolidated accounts, τους παγιωμένους λογαριασμούς και την επαναξιολόγηση όπου έχουμε και οδηγίες από ΕΕ. Τέλος, θεωρούμε ότι ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το θέμα της ανάπτυξης περαιτέρω προδιαγραφών και υποχρεώσεων benchmarks ώστε να είμαστε οι πιο υπεύθυνοι και να έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να είμαστε υπόδειγμα σε σχέση με την δράση επιχειρήσεων. Θα μπορούσε για παράδειγμα να υπάρξει η δυνατότητα να ασχοληθούν οι εταιρείε αυτές με το fair trade, το δίκαιο εμπόριο. Αυτά όσον αφορά και την ε, εθελοντική, το εθελοντικό σκέλο ε, τη ε, προσέγγισης, δεύτερο σκέλος, εξορθολογισμό. και οι βέλτιστες πρακτικές στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες στην ΕΚΕ, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτές οι δραστηριότητες, όμως γίνονται με ένα συντόνιστο τρόπο ουσιαστικά. Και έτσι είναι ανέφικτο για τους καταναλωτές, είναι αδύνατο οι καταναλωτές, το κοινό γενικά να κατανοήσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Εμείς θα ενθαρρύναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει δραστήρια αυτά τα θέματα και να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για βέλτιστες προδιαγραφές, benchmarking για αυτές τις ε, ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, ώστε να είναι πιο κατανοητέ, πιο εύληπτε και πιο συγκρίσιμε, καλύτερα συγκρίσιμε για του καταναλωτέ. Εκπονώντα ένα ενιαίο έγγραφο αναφορά, single document of reference, ώστε όσον αφορά τι ε, εταιρικά υπεύθυνε εταιρείε, ε, θα έπρεπε να ακολουθούν συγκεκριμένε ε, διατάξει και κατευθυντήριε γραμμέ και να βασίζονται στην υποχρέωση αυτή όσον αφορά τις, τα όσα απορρέουν από αυτή την προσέγγιση. Η συμμαχία ε, και ε, τα, ε, τα μέσα, τα εργαλεία αυτά είναι χρήσιμα, αλλά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε ένα input φιλόδοξο και αποτελεσματικό. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει οι απαντήσεις στην αγορά να έχουν μια υπεύθυνη συνιστόσα στην συγκυρία τους. Γιατί να μην υπάρξει η δυνατότητα indexing based human rights responsibilities, πρακτικών δηλαδή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ευθύνη για την τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα, Πρόεδρε, να αναφερθώ σε αυτό. Ένα τρίτο, μια τρίτη κατηγορία συστάσεων είναι ότι θα πρέπει να εξισορροπήσει, πιστεύουμε εμεί, την εξωτερική τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, επανισορροπώντα τα θέματα διαλόγου και λογοδοσία. Έχουμε την εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προφανώ μια προτεραιότητα όσον αφορά τι εξωτερικέ δράσει τη ΕΕ. Όμω επικεντρώνεται περισσότερο στο θέμα του διαλόγου. Το θέμα είναι δεν θα έπρεπε να ενταχθεί μέσα σε αυτή την προσέγγιση, σε αυτόν τον διάλογο πολύ περισσότερο το θέμα της λογοδοσίας για ε, τα θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα έπρεπε ως προς αυτό, για παράδειγμα, όχι μόνο να καλλιεργούμε διάλογο για να ξεπεράσουμε προβλήματα σε αυτά τα θέματα, αλλά να δούμε δυνατότητες και μέσα, εργαλεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί το capacity building, η δυνατότητα δηλαδή να είναι αποτελεσματικές οι τρίτες χώρες όσον αφορά την επιτήρηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την συμπεριφορά, την δράση εταιριών. Πιστεύουμε ότι ως προς αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα, όπως και στην αρχή της παρουσίασης αναφέρθηκε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εταιριών, της ευθύνη θα πρέπει να έχει ένα θέμα σε αυτόν τον διάλογο. Αυτή τη στιγμή η ο διάλογο επικεντρώνεται σε κρατικά προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι Τίθεται το ερώτημα, γιατί να μην ενταχθούν εδώ και οι εταιρείε, οι επιχειρήσει μέσα σε αυτόν τον διάλογο, ω ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου και έτσι να μπορεί μέσα σε ένα ανοιχτό διάλογο με κάθε ε, ε, ειλικρίνεια να συζητείτε Επίσης οι οικονομικές εταιρικέ σχέσεις και συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης είναι κάτι το οποίο εξετάζεται. Αυτό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται εδώ για να υπάρξει ένας μηχανισμός όρων και προϋποθέσεων ώστε να είναι πιο ελαστικό αυτό το πλαίσιο αυτών των μηχανισμών για να μπορεί να στοχεύουμε τις επιχειρήσεις με καλύτερο τρόπο. Έχουμε και μια κατηγορία τελευταία που απλά θα αναφέρω και δεν θα την επεξηγήσω θεωρούμε ευθυγραμμιζόμενοι με τις συστάσεις του ειδικού εντεταλμένου ότι ειδικά μέτρα επανόρθωσης είναι μία από τις πιο κέρυες πτυχές ε, της επιτυχούς πολιτικής ε, για τις εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούμε δεδομένη ε, της εμβέλειας και δεδομένων των δυνατοτήτων θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να υπάρχει λογοδοσία έναντι των θυμάτων και να υπάρχει μηχανισμός επανόρθωσης σε παγκόσμιο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάουτες. Να που ξοδεύονται καλά και τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογούμενων για μια φορά. Κύριε Μόρισον, εσείς είστε επικεφαλής του Ιστιντούτου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του κόσμου των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την, την Υποεπιτροπή για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια πρωτοβουλία που ιδρύθηκε το 2003 στις Βρυξέλλες και περιλαμβάνει οι εταιρείε που ηγούνται μια σειρά κλάδων με στόχο να δείξει πως η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων ανθρώπου μπορεί να ενταχθεί στην επιχειρηματική διοίκηση άσχετα από το γεωγραφικό χώρο, το πολιτικό πλαίσιο και, και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εμείς αναλάβαμε με μια προσέγγιση για να επιτρέψουμε και σε εμά και σε άλλες επιχειρήσεις να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό οι επιχειρήσει που μετέχουν σε εμά είναι από τι μεγαλύτερες στον κόσμο. ABB, Arriva, Barclays, Ericsson και πάρα πολλέ άλλε. Η πρωτοβουλία είναι υπό την προεδρία της Μέρι Ρόμπινσον, προέδρου στο παρελθόν της Ιρλανδίας και πρώην Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ. Αυτά που λέμε εδώ τα λέμε με αίσθηση ταπεινότητας. Οι εταιρείε που μετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή ξέρουν ότι είναι σύνθετο το ζήτημα, αλλά θέλουν να αναπτύξουν εμπιστοσύνη και προενεργή προσέγγιση στα δικαιώματα του ανθρώπου. Τα περασμένα έτη εξέτη ενίσχυσαν την πεποίθησή μας ότι φτάνουμε, περάσαμε την παιδική ηλικία, φτάνουμε σε μια άλλη κρίσιμη στιγμή στην ανάπτυξη, με μεγαλύτερη εμπλοκή κρατών και διακυβερνητικών οργανισμών. Κάποια από τα σχόλια που θα κάνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη. Και δεν, αποτελεί, δεν αποτελούν κριτική αλλά προς, πρόσκληση για συνεργασία. Έχουμε, είμαστε πρωτοπόροι στην υποστήριξη των από τις πλευράς επιχειρήσεων των εργασιών του κ. Ράγκη και την προστασία που, και το, της εργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης, αναφέρεται στο κοινό πλαίσιο και παραφέρεται ότι αποτελεί ένα καλό, καλά διαμορφωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του θεμάτων επιχειρήσεων και ανθρωπίνων και δικαιωμάτων που προωθεί σημαντικά τη συζήτηση. Αυτό το σχόλιο που, που τώρα δεν πρόκειται από τη Διεθνή Αμνηστία που θα μπορούσε να το κάνει αλλά από τρεις ε, επί... κύριε Μόλινσον δεν μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα θα Φοβάμαι για τον χρόνο, γι' αυτό μιλάω γρήγορα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό προέρχεται από τρει βασικέ ενό επιχειρήσεων. Τον Διεθνή Οργανισμό Επιχειρήσεων, τον, το Διεθνέ Εμπορικό Επιμελητήριο και την Συμβουλευτική Επιτροπή για τι Επιχειρήσει και τη Βιομηχανία, τον ΩΣΑ. Στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου θέλω να κάνω τρει παρατηρήσει. Πρώτον, οι επιχειρήσει χρειάζονται τα κράτη να υποστηρίξουν το κοινό αυτό πλαίσιο. Δεύτερον, η φύση τη συζήτηση εφελούσια ή υποχρεωτική, έχει υπερπολωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, υπάρχει πραγματική ευκαιρία να υπάρξει ευρωπαϊκή ηγεσία του ζητήματος. Και θα είμαι σύντομος. Πρώτον, οι επιχειρήσει χρειάζονται τα κράτη να υποστηρίξουν το κοινό πλαίσιο. Το, η κρατική υποχρέωση προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί από τι κυβερνήσει να παράσχουν ε, ισότιμο πεδίο, ε, ε, πεδίο λειτουργία για τι επιχειρήσει και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη νομοθεσία και σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ προσδοκίε. Βλέπουμε ότι συχνά οι επενδύσει, το εμπόριο, η εταιρική νομοθεσία πρέπει να ευθυγραμμιστεί περισσότερο και αυτό αυξάνει το, τη δουλειά των επιχειρήσεων κυρίως όταν το νομοθετικό πλαίσιο είναι και αντιφατικό. Χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των προσδοκιών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις και αυτών που ε, περιέχονται στις διμερείς εμπορικές και συμφωνίες, συμφωνίε, στι ε, συμφωνίες με τις κυβερνήσει των χωρών υποδοχή, στι ε, εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων και αλλού. Κάποια κράτη στην Ευρώπη έχουν αναλάβει ουσιαστική ηγεσία στο διάλογο με τις επιχειρήσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με άλλες περιοχές του κόσμου. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια πρέπει να αναλάβει ισχυρότερη θέση. Επίσης προσβλέπουμε στα κράτη για να ε, επιβάλλουν να λογοδοτούν οι τζαμπατζίδες, οι αυτοί που καθυστερούν και να δώσουν να υπάρξει μεγάλη, καλύτερος μηχανισμός λογοδοσίας αυτών που πλήττουν τις επιχειρήσεις χωρίς να κάνουν τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ενισχύσει τα εθνικά σημεία επαφής του ΩΣΑ και να βοηθήσει τη δημιουργία ενός ombudsman, στην, ενός διαμεσολαβητή στην Ένωση. Επίσης, είναι κρίσιμο να εμπλακούν στις συζητήσεις και άλλες περιφέρειες, ώστε οι επιχειρήσεις από την Αφρική, την Ασία και την Αμερικανική Ήπειρο να ελέγχονται και αυτές από τις κυβερνήσεις τους. Αυτή τη στιγμή κάποιες λίγες ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ε, προσελκύουν ε, ένα μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας του κοινού για τη συμπεριφορά του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικές φορές αυτό ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αλλά Άλλες φορές κρύβεται, αυτό κρύβει την, την ανάγκη να ελέγχονται επιχειρήσεις από την Κίνα, τη Ρωσία, τη Βραζιλία και την Ινδία που είναι πολύ πιο υπεύθυνε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρώπη ωστόσο θα μπορούσε σίγουρα να λειτουργήσει σαν παράδειγμα και εμείς μπορούμε πολλά ακόμα να κάνουμε για να παίξουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε έναν πρωτοπόρο ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης τα κράτη ε, μπορούν να παίξουν και άλλο ρόλο σε κρατικές ή μη κρατικές επιχειρήσεις. Έναν άλλο τομέα στον οποίο μπορούν να παίξουν τα κράτη είναι όταν κάποιες επιχειρήσεις είναι βασικές, βασικοί προμηθευτές των κρατών. Όταν υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν ε, ανάγκη, δεν έχουν επαρκή δυνατότητα και χρειάζονται κοινές, κοινούς πόρους. Επίσης, κάποιες επιχειρήσεις που μπορεί να μην και εισηγμένες στις ε, άκρες της Ευρώπης να, να είναι λιγότερο υπόλογες. Αυτό πρέπει να διορθώσει. Να διορθωθεί. Δεύτερο θέμα. Όπως σας είπα έχει γίνει μια υπερβολική πόλωση ανάμεσα στο αν πρέπει το πλαίσιο να είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό. Το, οι, προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις επιχειρήσεις είναι σύνθετα διλήμματα σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη δεν μπορούν να προστατεύσουν τον πληθυσμό λόγω σειράξεων, διαφθοράς, φτώχειας. Υπάρχει άνισο επιχειρηματικό καθονιστικό περιβάλλον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι επιχειρήσεις συχνά πρέπει να λύσουν και ζητήματα που αφορούν στον πληθυσμό και ζητήματα που αφορούν τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη, αλλά συχνά οι επιχειρήσει βρίσκονται μπλεγμένες ανάμεσα στις επιχειρηματικέ προσδοκίες μιας επιχείρησης και τις απαιτήσει για ανθρώπινα δικαιώματα κρατών και περιφερειών. Μια προσέγγιση της εταιρική ευθύνη, τη ε, της κοινωνική κοινωνικής με νόημα στα 27 κράτη θα ήταν να υπάρχει ένα, ένα ε, ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι καλό, αλλά σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό δεν έχει νόημα όταν λειτουργούν επιχειρήσει έξω από την Ένωση. Τελευταία παρατήρηση. Υπάρχει πραγματική ευκαιρία να αναλάβει την ηγεσία η Ευρώπη. Κάποιες από τις καλύτερες ε, συνεργασίες ε, κυβερνήσεων και επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγιναν εκτός Ένωσης. Και συχνά όταν ενεπλάκησαν ε, κράτη τη Ευρώπη, αυτό έγινε μάλλον παρά παρά χάρη στην ευρωπαϊκή εμπλοκή. Κάποιε από αυτέ ε, ε, συνεχίζονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ασία. Οι επιχειρήσεις θέλουν, είναι πρόθυμες να αναλάβουν ηγετικέ θέσει στα δικαιώματα των εργατών, στι αλυσίδε προμήθεια, στον τομέα της ασφάλειας, του, της επιχειρήσης πετρελαίου και της εξωτική. Ε, ε, και τις εξωτικές βιομηχανίες. Τώρα έχει πολλές πλευρές, από το Google και το Yahoo μέχρι το ότι η Novartis ε, ε, και οι Novo Nordisk αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην υγεία, ενώ η Suez, η Thames, η Water, η Coca-Cola και η Pepsi αναγνώρισαν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την κατοχή του νερού. Χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με αυτό τη ηγετική θέση των επιχειρήσεων. Γιατί και αυτό θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στο πλαίσιο του κυρίου Ράγκη. Εμείς ε, ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει το πλαίσιο αυτό και να εμπνεύσει και τις δικές σας και τις δικές μας δράσεις τους επόμενους μήνες και τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Καζάλς, ως συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Δικαιοσύνη στις Επιχειρήσεις, με Πολλέ ΜΚΟ που είναι και αυτοί που εκπροσωπούνται κυρίω στην αίθουσα. Έχετε να μα δείξετε κάτι κύριε Καζάλη. Ça va marcher.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 Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Υποεπιτροπή για την μεγάλη ευκαιρία που μας δώσετε σήμερα να είμαστε παρόντες. Εμείς ετοιμάσαμε ένα έγγραφο ειδικά για αυτή την ακρόαση. Είναι στην είσοδο, είναι από πολλές οργανώσεις και είναι μια σύνοψη αυτό που θα σας πω τώρα. Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός ECCJ είναι α, α, καλύπτει 250 περίπου ε, οργανώσεις για το περιβάλλον, συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, από όλο τον κόσμο όπως η Διεθνή Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και εθνικά τμήματα της ε, Διεθνούς Αμνηστίας, Oxfam, Greenpeace και πολλά άλλα. Για αυτή εδώ την ακρόαση συνεργασία με την ΚΑΦΟ το Βέλγιο, Ολλανδία, δράση στην Ολλανδία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ισουητών στις Βρυξέλλες και το Global Witness. Θα αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, η κατανόηση του τι εμείς θεωρούμε πρόβλημα και τι κάνουμε. Καταρχήν το νομικό σύστημα δυσλειτουργεί και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι πολιτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την ευθύνη που θα έπρεπε έναντι της κοινωνίας. Έχουμε ατιμορρησία και έλλειψη μέσων διόρθωσης που επηρεάζουν κυβερνήσεις, ε, κοινότητε και άτομα που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης για νομική θεραπεία των πληγμάτων τα οποία υπέστησαν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Μερικές ε, ε, επιχειρήσεις ε, εποφελούνται από την ενιαία αγορά, άλλες δεν εποφελούνται όσα θα έπρεπε. Επειδή οι πρώτες κάνουν κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μιλάω κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι θα έπρεπε να γίνει και γι' αυτό. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το Κονγκό. Η Global Witness μας έδωσε τα στοιχεία. Έχουμε μια βρετανική εταιρεία, Aframex, το Φεβράριο του 2007, η Global Witness κατέγγειλε την εταιρεία Aframex για το ότι δεν τηρούνται οι κατευθυντήρες γραμμές για τις επιχειρήσεις. Έγινε μια έρευνα και τον Αύγουστο του 2008 δημοσιεύτηκε το πόρισμα που επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της Global Witness και έγιναν συστάσεις προς την Αφρομέξ κυρίως για την εφαρμογή και περιοδική αναθεώρηση ε, πολιτικής εταιρικής ευθύνη που θα λαμβάνει υπόψη την επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρασαν εννέα μήνες από το πόρισμα. Ακόμα δεν έχει φτάσει πληροφορία από την εφημερίδα για το πώς εφάρμοσε τις συστάσεις. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το Κονγκό. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Και όλα μας δείχνουν τα προαιρετικοί, ή προαιρετικοί μηχανισμοί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δίνουν λύση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι κατευθύνες γραμμές της, του ΟΣΑ ήταν προαιρετικές. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια πιο δεσμευτική μέθοδος. Όπως είπε ήδη το Ευρωκοινοβούλιο και άλλοι σημαντικοί όπως η G8, τα προαιρετικά μέτρα δεν είναι και δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν νομοθεσία όπου αυτό επιβάλλεται. Δεύτερο θέμα για σήμερα. Η Ένωση πρέπει να δράσει. Το πλαίσιο που παρουσίασε ο καθηγητής Ράγκη δίνει γόνιμο έδαφος στην Ένωση και στη διεθνή κοινότητα να στηριχτεί και να προχωρήσει. Δίνει μια ιστορική ευκαιρία για την Ένωση, για δράση. Ελπίζουμε ότι η Ένωση και ο καθηγητής Ράγκη θα συνεργαστούν για να έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνες γραμμές του τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να βελτιώσουν την, το χαρακτήρα υπολογίας των επιχειρήσεών τους. Θεωρούμε ότι θέματα όπως η ευθύνη των χωρών, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι σημεία κλειδιά. Εμείς θα συνεργαστούμε γι' αυτό και με τον καθηγητή και με την Ένωση. Χωρίς τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την πρόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία της βιοδιαφορετικότητας, τη δημιουργία απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, αυτά όλα δεν γίνονται αν δεν δει η Ένωση τι κάνουν οι επιχειρήσεις της και τι κανόνες ισχύουν και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Ζούμε με οικονομική κρίση μεγάλη. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ξανασκέφτονται τα πράγματα. Ξαφνικά οι ε, κανονισμοί ο όρος κανονισμός έχασε μια κακή χρειά που είχε ως έννοια. Βλέπουμε ότι η Κομισιόν άρχισε να ακούει σιγά σιγά τις θέσεις μας. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου ήταν πολύ σημαντικός για αυτή την αλλαγή στάσης και λόγω της πίεσής μας λοιπόν και μια, μια μελέτη που θα γίνει από τη Γενική Διεύθυνση για τις Επιχειρήσεις όπου θα ορίζονται πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις ευθύνες των επιχειρήσεων της Ένωσης στη δράση του στο εξωτερικό. Οπότε σιγά σιγά η Κομισιόν καλό θα είναι να τη δοθεί μια πιο ευρία εντολή να εντοπίσει τα προβλήματα και να τα εντοπίσει όπου χρειάζεται. Ο καθηγητής Βόλτερς ε, σωστά έθεσε το θέμα στη σωστή του διάσταση που είναι η, διάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτο πεδίο, τι δουλειά κάναμε εμείς ως μη κυβερνικές οργανώσεις και τι λύσεις προτείνουμε. Μία μελέτη που σας παρουσιάσαμε τον Μάιο πέρυσι και είναι και αυτό στην είσοδο της αίθουσας και στην ιστοσελίδα μας αναφέρει τρεις δυνητικές λύσεις. τις οποίες προσπαθούμε να τις βελτιώνουμε. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις Συνήθως είναι πολλά χωριστά νομικά πρόσωπα. Αυτό περιορίζει και την ευθύνη τους κατά κάποιο τρόπο. Έπειτα οι μητρικές εταιρείε και οι διευθυντές κατά κάποιο τρόπο προστατεύονται να μην είναι υπεύθυνοι γιατί το τι ε, δυσλειτουργίες συμφωνίζονται μέσω των υπεργολάβων κλπ. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν το δάγμα της περιορισμένης ευθύνης. Τι εννοώ και τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, στο slide αυτό, μία μητρική εταιρεία στην Ευρώπη ωφελείται από διάφορες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η ευθύνη είναι πολύ πιο κάτω στο επίπεδο της αλυσίδας. Εμείς θέλουμε οι μητρικές εταιρείες μέσω κανονισμού να είναι υπεύθυνε για παραβιάσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον κλπ. Επίσης, οι διευθυντές και οι μητρικές εταιρείε θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα ο νόμος να ασκεί ανακρίσει σε βάρος τους στα πλαίσια της ευθύνης τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ενεργό, ενεργής υποχρέωσης φροντίδος φροντίδας, diligence όπως το χαρακτηρίζει ο καθηγητής Ράγκη, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό. Uh, Άλλο θέμα είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τι νόημα έχει να υπάρχει νομοθεσία αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί εφαρμογής. Η αποτελεσματικότητα ενό κανονισμού εξαρτάται από την πόσο εφαρμόσιμος είναι. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κάθε πολίτης να φέρει, να κάνει μια ε, προσφυγή σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση που υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει η αποζημίωση, το βάρος της ε, απόδειξης της ευθύνης και διάφορα άλλα νομικά εμπόδια που σήμερα υπάρχουν να αρθούν. Οι μη κυβερνικέ οργανώσεις επίσης θα πρέπει να έχουν πιο σαφή θέση μέσα στο πεδίο, στο όλο πεδίο προκειμένου να προωθούνται αυτά τα αιτήματα. Το τελευταίο θέμα αφορά διαφάνεια και τα συναφή. Όπως είπε και ο καθηγητής Γότερς και το, το έχετε πει πολλές φορές στο κοινοβούλιο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που λειτουργούν ιδιαίτερα στην αγορά της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν συγκρίσιμες ε, προδιαγραφές, μη οικονομικές εννοώ. Να στηριχθούμε στις βέλτιστες πρακτικές, να μην ξεκινήσουμε από το μηδέν. Υπάρχει ήδη ένα δεδομένο, μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό. Υπάρχει ήδη νομοθεσία της Ένωσης. Το σημαντικό είναι η έκθεση αυτή να έχει πρώτον την ταυτοποίηση της ομάδας επιχείρησης και ποια είναι το πεδίο ευθύνης μιας εταιρείας. Να ορίσει τι κίνδυνοι υπάρχουν για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι μπορεί να κάνει η επιχείρηση γι' αυτό και τρίτο ποια είναι η επίπτωση συγκεκριμένη στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πεδίο ευθύνης της εταιρείας. θα πρέπει να υπάρχουν κλαδικοί ή τομεακοί μάλλον δείκτες Δεν μπορεί αυτό να εφαρμόζεται γενικά για όλους τους κλάδους και τομείς. Οι διευθυντές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την έκθεση αυτή και να έχουν και την τελική ευθύνη στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα. Θέλουμε οι μη κυβερνικές οργανώσεις και τα πληττόμενοι πολίτες και θύματα να έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν σε δικαστήριο κατά τις εταιρεία, πράγμα το οποίο δεν γίνεται σήμερα υπάρχει και ανεξάρτητος έλεγχος για την επιβεβαίωση της ε, αληθείας των στοιχείων της έκθεσης. Μπορούν οι προτάσει αυτέ να καλυφθούν σε ένα βαθμό με τροπολογίε τη νομοθεσία που ήδη υπάρχει, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να μα βοηθήσει σε αυτό. Και τελειώνω με το εξή. Με συστάσει προτάσεις προς το Ευρωκοινοβούλιο. Έχω μια μεγάλη ευκαιρία τις ευρωεκλογές σε δύο μήνες. Ελπίζουμε οι πολιτικές ομάδες να συμπεριλάβουν μερικά από τα αιτήματα αυτά για την ευθύνη των επιχειρήσεων στο εκλογικό τους πρόγραμμα. μας χάρη στη Γαλλία έχει γίνει αυτό ήδη σε έναν βαθμό. Δεύτερο, μετά τις ευρωεκλογέ το Κοινοβούλιο, ένας από τους σημαντικούς του ρόλους, θα είναι να δώσει το πράσινο φως στη νέα Κομισιόν. Θα θέλαμε οι αρμόδιες επιτροπές να δούνε το θέμα αυτό πάρα πολύ καλά, η μυρίσια διάταξη ευθύνης των επιχειρήσεων σε κάθε, ε, κάθε επιτροπή σε σχέση με την Κομισιόν. Επίσης θέλουμε στο μέλλον περισσότερες συζητήσεις για την ευθύνη των επιχειρήσεων σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Συνήθως η Επιτροπή Αποσχόλησης το κάνει. Έχουμε και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες επιτροπές που θα έπρεπε να παίρνουν μέρος στη διεργασία αυτή, να καλούν θύματα κλπ. Το Κοινοβούλιο επίσης θα πρέπει να διασφαλίσει με βάση μια γενική διεύθυνση της Γενική Διεύθυνση των Επιχειρήσεων όρισε να καθοριστεί το πλαίσιο όσον αφορά την κοινωτική νομοθεσία. Τι ισχύει για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πού υπάρχουν κενά. Τι δυνατότητες υπάρχουν για περαιτέρω δράση. Ελπίζουμε σε αυτό να παίξει ρόλο και το Κοινοβούλιο. Έπειτα έχετε δημοσιονομικές εξουσίες. Ήδη υπάρχουν προγράμματα για επιχειρήσεις που θα πάρουν χρήματα για αναπτυξιακά προγράμματα ή σε αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ κριτήριο όσον αφορά τα ανθρώπινα κριτήρια. Αυτά πρέπει να τα κάνει το κοινό. Για την Ένωση πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη συνεργαζόμαστε με τον καθηγητή Waters ή θα συνεργαστούμε κι άλλο αν ενδιαφέρεται για προτάσεις. Υπάρχουν όμως τρία κομβικά σημεία που πρέπει να τα δούμε. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρχει μια δήλωση του Συμβουλίου ή κάποια διακήρυξη τέλο πάντων που να αναγνωρίζει το ότι υπάρχει το, ένα διεθνές πλαίσιο όπως προτάθηκε από τον και γνωρίζει τις ευθύνες των κυβερνήσεων και των εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον τρόπο θεραπείας των προβλημάτων. Πρέπει να δοθεί συνέχεια στη μελέτη της Κομισιόν όπως είπα και τρίτο, ένα πρώτο βήμα θα πρέπει να οριστούν οι ευθύνε. Ποιο είναι υπεύθυνο για αυτά στι υπηρεσίε τη Κομισιόν, γιατί τη στιγμή υπάρχει ασάφεια. Ποιο είναι υπεύθυνο για την εταιρική ευθύνη. Δεν υπάρχει ένα υπεύθυνο σε επίπεδο ενό Ο καθηγητής Ράγκη είπε ότι μερικές χώρες ήδη έχουν τμήματα υπηρεσίες γι' αυτό. Αυτό δεν συμβαίνει στην Κομισιόν. Να ξεκαθαρίσει λοιπόν ποιος έχει ποια ευθύνη και να δοθούν και περισσότερα κονδύλια. Αυτά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Καζάλ καλά δουλέψατε στην συντονιστική σας ομάδα με ένα ωραίο πρόγραμμα δράσης. Σας υπενθυμίζω ότι και στην έκθεση της κυρώσης που ήταν μία από τις πρώτες ε, τέσσερις ε, εκθέσεις της Επιτροπής επιβάλαμε στο Κοινοβούλιο να ζητήσαμε το Κοινοβούλιο να επιβάλλονται κυρώσεις στις επιχειρήσεις και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για παραβίαση του δικαιώματος των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, κάτι που υποστήριξε το Συμβούλιο στην Ολομέρεια στη συζήτηση. Πρόκειται για ένα τομέα που και εμένα με βρίσκει σύμφωνη, χωρί κυρώσει. είτε μέσω της διεθνούς δικαιοσύνης είτε μέσω της ε, ευρωπαϊκή ε, της ευρωπαϊκής ε, δικαιοσύνης είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση περνάει κάποια βασικά θέματα. Τελευταίο εισηγητής ο κύριο Εύανς, επικεφαλή, της, συμβουλευτική της επιτροπή των ΩΣΑ και δουλέψατε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, είμαι υπεύθυνο τη ΤΟΑΚ αλλά συνεργαζόμαστε και με την ETUC και άλλες κλαδικές ομοσπονδίες συνδικάτων. Ήθελα σήμερα να σας δώσω κάποιες προσωπικές απόψεις και για το πλαίσιο τη συζήτηση ε, του έργου του κύριου Ράγκη και για την εμπειρία που είχαμε χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο, τις οδηγίες του ΩΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις τα τελευταία 8 χρόνια όπως ξέρετε άλλαξαν σημαντικά το 2000. Στο πλαίσιο, για το πλαίσιο τώρα. Η σημασία των συζητήσεων για τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ των μελών μας. Στον ιδιωτικό τομέα τα περισσότερα μέλη μας δουλεύουν σε κάποια μορφή αλυσίδα και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ε, μείωση των δυνατοτήτων που είχαμε. Αλλάζει η σχέση ε, δυνάμεων στο παρελθόν. Μπαίνει ωστόσο και το γενικότερο ζήτημα της λογοδοσίας των επιχειρήσεων. Δεύτερον, τα μέλη μας αναζητούν πρακτικές λύσεις για να επιλύσουν κάποια από τα ζητήματα που ανακύπτουν και να αυξηθεί ο, ο χώρος, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία σε διεθνές επίπεδο και με τις κυ... κυβερνητικές δομές. Άκουσα αλλού να λέει ο κύριος Ράγκη ε, να περιγράφει τις ε, συζητήσεις στη Γενέβη ως ένα σειροδρομικό ε, ναυάγιο. Ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε της, ε, το κίνδυνο σύγκρουσης. Τα τελευταία χρόνια στις συζητήσει για την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Κομισιόν μιλάγαν όλοι για προ, προαιρετικό ρόλο. Και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή αντί να προχωρήσει προς τα μπρος προχώρησε προς τα πίσω. Και όπως τόνισε και σήμερα ο κύριος Ράγκη οδήγησε σε κινησία τους μεγαλύτερους εμπλεκόμενους στον τομέα. Άρα πρέπει να φύγουμε από αυτό το αδίέξοδο. Όπως αναφέρθηκε επίσης πριν από λίγο, η συζήτηση γίνεται στα πλαίσια της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι συζητήσεις για την αλλαγή του κλίματος περιγράφηκαν πριν από δύο χρόνια ως η μεγαλύτερη εμπορική αποτυχία στην ιστορία από κάποιους οικονομολόγους. Φέτος νομίζω ότι φέτος και πέρσι η οικονομική κρίση παίρνει τα ενία. Και είναι σαφές ότι η αυτορύθμιση σε πολλές περιπτώσεις σημαίνει μη ρύθμιση. Και η συνέπεια για την, το αν η εταιρική ευθύνη είναι προαιρετική ή υποχρεωτική ανατρέπει τις συζητήσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο. Εάν η Γενέβη ήταν ένα μια σύγκρουση τρένων. Τώρα έχουμε μπροστά μας πολλά, πολλές δυνητικές συγκρούσεις μεταξύ κυβερνήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ αγορών που θα έχουν συνέπειες και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με δεδομένο το πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για το πλαίσιο του κυρίου Ράγκη. Protect, Respect, Remedy. Το κείμενο όντως επιτρέπει να προχωρήσουμε αναζητώντας πρακτικές λύσεις σε κάποιο από τα ζητήματα. Πρώτον, για την εμπειρία που είχαμε σε ό,τι αφορά την κρατική υποχρέωση, το κρατικό καθήκον προστασίας. Ένα, το βασικό πρόβλημα, σωστά το τονίζει η έκθεση Ράγκη, η θεσμική δυσλειτουργία στο εσωτερικό των κυβερνήσεων, που εμφανίζεται ακόμα εντονότερα σε διεθνές επίπεδο. Πώς οι κυβερνήσεις ασκούν συνεκτικές πολιτικές. Αυτό δεν αφορά μόνο τον τομέα εκτός των εργασιακών ε, προδιαγραφών και εδώ θα διαφωνήσω λίγο με αυτά που είπε ο κύριος Ράγκη γιατί μας είπε ότι υπάρχει στον παγκόσμιο, στο Παγκόσμιο Γραφείο Εργασίας υπάρχει μια διαδικασία που δουλεύει, ενώ σε άλλους τομεί όχι. Αυτό όντω είναι σωστό σε ό,τι αφορά νομολογία, εντοπισμό ζητημάτων και οι οδηγίε του ΩΣΑ στηρίζονται σε αυτά τα στάνταρ του διεθνού Γραφείου Εργασίας. Ωστόσο, η εφαρμογή του χωλαίνει ακόμα και υπάρχει μια δυσλειτουργία μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων των κυβερνήσεων όπω αντικατοπτρίζονται στους δεσμευτικούς κανονισμούς που υπάρχουν στις επενδυτικές συμφωνίες ή στις εμπορικές συμφωνίες και την ρυθμιστική προσέγγιση των ε, εργασιακών δικαιωμάτων. Άρα, για μας, εμείς θεωρούμε ότι η εφαρμογή των ε, οδηγιών του ΟΣΑ ε, στον τομέα των δικαιωμάτων είναι πολύ χαλαρότερη από αυτήν που βλέπουμε στις εμπορικές συμφωνίες, στις συμφωνίες διαιτησίες ή στην εφαρμογή της αστικής νομοθεσίας σε πολλούς τομείς. Η αναθεώρηση των οδηγιών αυτό του 2010 ε, είναι ένα σημαντικός παράγοντας, αλλά θα ήθελα να πω ότι η βασική... Το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει εξισορρόπηση σε σχέση με τα θέματα εξουσιών όσον αφορά τα θέματα κοινωνικών προδιαγραφών μέσα στο έργο αυτό δείξαμε πλευρά συνδικάτων παράλληλα με περιπτώσεις ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και στις περιπτώσεις DRC 100 περιπτώσεις όσον αφορά εργασιακές προδιαγραφές ε, από το 2001 και την αναθεώρηση. Εξετάσαμε τις επιπτώσεις και το ίμιση περίπου ολοκληρώθηκε ή επιλύθηκε με τον ένα ή άλλο τρόπο από τις 50 περίπου 25 επιλήθηκαν με έναν τρόπο που ήταν θετικό σε σχέση με την εναλλακτική λύση που θα ήταν α, η άλλη επιλογή όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από τις 25-12 περίπου το ίμιση έχουν αναφερθεί όσον αφορά την ε, κομβική ε, υπηρεσία, όσον αφορά την παρέμβαση του κράτους για να υπάρξει επίλυση. Πολιτική ευθύνη ή πολιτική βούληση λείπει κατά την άποψή μου. Επίσης, συζητήσεις για θέματα εξάρτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με άλλες συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες. Όντως πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των προσδοκιών των κρατών ως καλή συμπεριφορά από τις επιχειρήσεις και το τι είναι έτοιμες να υποστηρίξουν οικονομικά. Και οι επιχειρήσεις λένε «Α, αυτό δεν στέκει γιατί αυτό αλλάζει το προαιρετικό και το κάνει υποχρεωτικό». Βεβαίω, δεν είσαι υποχρεωμένο να πάρει κρατικά κονδύλια. Αν δεν θε, τα παίρνει. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Και, ωστόσο, το ζήτημα αυτό μπαίνει στο κέντρο τη συζητήσεων γιατί με αυτόν τον τρόπο η αύξηση των εξαγωγικών πιστώσεων από τι κυβερνήσει χωρίς σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργεί ανισότητες. Είναι λοιπόν τομέα στον οποίο και οι κυβερνήσει θα μπορούσαν να ε, προχωρήσουν. Συγγνώμη που πάω γρήγορα, ξέρετε, κουλτικό είναι. Να μπω στο θέμα των δυνατοτήτων προσφυγής και των νομικών θεραπείων. Προφανώς σημαντικός ρόλος σε εμάς είναι τα εθνικά σημεία επαφής. Και εδώ ωστόσο οι υπηρεσίες μας λένε ότι το ίμιση έως και τα δύο τρίτα των εθνικών σημείων επαφής λειτουργούν όπως ε, προσδοκάται με διαμεσολάβηση και με παρεμβάσεις. Κάποια θετικά αποτελέσματα είναι, υπάρχουν, αλλά περιορισμένα. Στη Βρετανία το Εθνικό Σημείο Επαφής έκανε μια διαμεσολάβηση επιτυχή μεταξύ ε, συνδικάτων και μιας επιχείρησης. Υπάρχει το θέμα όμως του πού βρίσκεται το Εθνικό Σημείο Επαφής στο Υπουργείο Οικονομίας ας πούμε για τους εμπλεκόμενους δεν είναι ε, καθοριστικό και θεωρείται χαμηλής προτεραιότητας. Εξαρτάται από το αν είναι διμερής, τριμερής ή τετραμερής η η διαμεσολάβηση. Αν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει συνέχιση παρουσίας του προσωπικού, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε πόδους. Η καλή πρακτική στην πράξη είναι εξαίρεση, όχι κανόνας. Ίσως να κλείνετε κύριε Evans. Έλεγα για να κλείσω τι γίνεται σε σχέση με την κρίση. Βρισκόμαστε, κάποια θέματα είναι σε σταυροδρόμι. Από τη μια μεριά, η οικονομική πίεση προς τις επιχειρήσεις και η ανάγκη περικοπής δαπανών οδηγεί σε περικοπές ακόμα και προσπαθειών να περάσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη μπροστά. Από την άλλη μεριά, οι κυβερνήσεις ελέγχουν μεγάλο τμήμα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και το θέμα της μελλοντικής διαμόρφωσης του σκηνικού πέφτει στα χέρια τους. Στα χέρια τους. Στις συζητήσεις του G8 και του G20 είχαν γίνει κάποιες προτάσεις από, τον Μέρκη, από τη Μέρκη και από τον Τρεμόντι για το πώς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Τελευταία τελευταία συνάντησή μας είναι αυτή. Πάλι δεν είχαμε πολύ χρόνο. Δεν ζητώ από τους συναδέλφους αν θέλουν να λάβουν το λόγο γιατί και αυτό είναι πραγματικά δραματικό. Έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Η Άννα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τους εισηγητές τους ομιλητές σημαντικότατη πρωτοβουλία. Να τονίσω ότι αυτό απαιτεί κοινή δουλειά πολλών επιχειρήσεων, πολλών επιτροπών συγγνώμη, του Κοινοβουλίου στην επόμενη θητεία. Όπως προτείνουν η ΜΚΙΟ. πολλά από αυτά τα εφαρμόζουμε ήδη ή τα προσπαθούμε να τα περάσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Ω αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλοί βουλευτές, ανεξάρτητα από το κόμμα και την εθνική καταγωγή, ξεκίνησαν μία αναφορά και αν θέλετε να την υπογράψετε για να τη διαδώσετε, για να σταματήσει η διαφθορά. Και η ερώτησή μου προς τον κύριο Ράγκια είναι ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους μηχανισμούς νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς ώστε να συνεργάζονται με τους μηχανισμούς ε, που θέλετε να δημιουργήσετε για την ε, προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπου. Γιατί συχνά οι επιχειρήσει που, που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε τρίτε χώρε είναι, είναι εκείνε που ασχολούνται και με την διαφθορά υπαλλήλων, την Ε, κατά την ε, υπεξαίρεση πόρων από την ανάπτυξη που είναι στην ουσία παραβίαση δικαιωμάτων, ε, βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Δεν θα ήταν αποτελεσματικότερο να συνδέσουμε τις δύο αυτές διαστάσεις και να ζητήσουμε. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ένωση αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ την Αναγκούμες. Η Βερονίκ Δεκάιζερ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα απαντηθεί. Μπήκε ο κύριος Εύαν σε αυτό που ήθελα να πω. Ευχαριστώ τους συζητητές παρεμπιπτόντως. Είπε ο κύριος Εύανς ότι οι νέες δομές που θα τεθούν σε ισχύ δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο που μπορεί να αλλάξει τι θα συμβεί εν ώψη της οικονομικής κρίσης. Όχι μόνο της χρηματοεπιστοτικής κρίσης, αλλά και της οικονομικής κρίσης. Ο κ. Σεβάνς απάντησε εν μέρη. Λέμε, ο νέος ρόλος των κυβερνήσεων στην ε, ενίσχυση, στις ενισχύσεις που χορηγούν και τη δυνατότητα να εξαρτηθούν οι ενισχύσεις με κάποια μορφή σεβασμού του περιβάλλοντος κλπ. Μικρή απάντηση Ωστόσο, αν δεν έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις θα κάνουν προσπάθειες. Βρισκόμαστε σε μια σύνθετη κατάσταση και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της νέας φοιτίας, πρόεδρε, όπου ελπίζω να σας ξαναβρω εδώ, πρόεδρε, ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε τη συζήτηση στο νέο πλαίσιο. Γιατί θα χρειαστεί να το κάνουν ούτως ή άλλως δεδομένων των μηνών και ετών που μας αναμένουν. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό, στηριζόμενοι ακριβώς σε αυτό το νέο πλαίσιο. Δεν περίμενα απάντηση βέβαια τώρα. Θα ζητήσω από τον κύριο Χάουιτ να θέσει την ερώτηση που θέλει να θέσει και να δώσει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Όλοι βλέπουμε ότι αυτό είναι θέμα προτεραιότητας για την επόμενη θητεία θα το δουλέψεις, οπότε ενδεχόμενα θα μπορέσεις να προσανατολίσεις τις συζητήσεις για το μελλοντικό κοινοβούλιο. Και μετά θα μας τα πει συνοπτικά. Σύντομα, γιατί ήδη έχουμε πάει στους παρα 25. Um, σας ευχαριστώ. Θα ερμηνεύσω την ερώτηση πολύ στενά και συνοψίζω λοιπόν επειδή δεν έχουμε χρόνο. Έχω δύο ερωτήσει προ τον Τζον καταρχήν. Πρώτα σε ευχαριστώ για αυτό που είπες. Για τη διαφορά μεταξύ προαιρετικών και υποχρεωτικών. Δεν θέλω να επαναλάβει αυτό. Σε ευχαριστώ που έκανε αυτή τη διάκριση στους ορισμού. Αλλά κάτι από αυτό που κάνεις στην Γενέβη είναι εξασφάλισε αυτή την υποστήριξη. Σε συγχαίρω γι' αυτό. Πώς το κατάφερες. Δεν λέω ότι μπορούμε εμείς να επαναλάβουμε εδώ, μπορούμε να διδαχτούμε. Πώς το κατάφερες το έργο αυτό στη Γενέβη. Και δεύτερον, σε σχέση με αυτά που είπε η Στάφος Βερονίκ Ντικέζερ για την κρίση που ζούμε. Είπε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία γι' αυτό. Τα πράγματα να αλλάξουν, να προωθηθεί η υπόθεση αυτή. Αλλά για να πω και το αντίθετο, εγώ ανησυχώ. Επειδή έχουμε ένα τεράστιο οικονομικό χρηματοπιστωτικό πρόβλημα, οι κυβερνήσει να το ερμηνεύσουν χρηματοπιστωτικά και να στήσουν ένα σωρό νέε υποχρεώσεις αναφορών κλπ. Αλλά μόνο με στενά χρηματοπιστωτικά κριτήρια. Και μετά από 10 χρόνια να διαπιστώσουμε ότι χάσαμε μία δεκαετία. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Και τέλος, σε σχέση με αυτό που είπες εσύ, Ελέν, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για απάντηση από την Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν έχει κανένα λόγο να απολογείται. Εξ ονόματος, για μάλλον της Κομισιόν, λέω ότι όλα αυτά που ακούστηκαν δεν είναι επικρίσεις, είναι και πολλά επενετικά σχόλια. Πάντως δεν έχουμε αρκετή ηγετική φυσιογνωμία στο θέμα αυτό από την πλευρά σας. Και αυτό είναι σωστή κριτική. Και θέλω να μαρτυρήσω ότι η μελέτη που έχει ορίσει να γίνει η Κομισιόν για την υποχρέωση των επιχειρήσεων μπορεί να στηριχθεί στη δουλειά του Τζον, δεν υπάρχει λόγος να επαναφευρίσκουμε τον τροχό, αλλά μπορεί και να συμβάλλει στην εντολή του το 2011. Αν το κάνουμε αυτό, θα επιδείξουμε ηγετικό ρόλο. Έχετε δεσμευτεί γι' αυτό. Και το λέω δημοσία. Σας πιστώνω με αυτό. Αν υπάρχει μια ευκαιρία και χρόνος για απάντηση της Κομισιόν, ίσως κάποια από την Γενική Διεύθυνση για τις Εξωτερικές Σχέσεις, διευθύνσεις μάλλον, Πώς εξασφαλίζετε αυτή τη συνοχή, μήπω απλώ ψηφίσατε στη Γενέβη και μετά ξεχάσετε τι ψηφίσετε ή τα εφαρμόζετε κιόλα. Όχι όπω κάνουν οι κυβερνήσεις, αλλά όπω κάνουμε συλλογικά στην Ένωση με τα προγράμματά μας. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει με προσοχή να παρακολουθήσουμε από εδώ και μπρο και μετά τι ευρωεκλογέ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε σα, Κύριε Ράγκη πολύ σύντομα σας παρακαλώ δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο τα πορίσματά σας, τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ σύντομα θα απαντήσω σε ερωτήσεις και μετά θα μπορέσουν οι δόλοι διερμηνείς να πάνε και να γευματίσουν. Σύνδεση με την διαφθορά. Αυτό σε σχέση η διαφθορά για την επίτευξη της, ε, των στόχων μας είναι κίνδυνος. Όμως δυστυχώς όπως και αν το δει κανείς, η εντολή μου ρητά αποκλείει το να εξεταστούν θέματα διαφθοράς, διότι υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που λειτουργούν γι' αυτό ξεκινώντας ε, με, την, με τον νόμο για τις ε, ε, πράξεις στην αλλοδαπή όσον αφορά διαφθορά έχει και την σύμβαση των Ηνωμένων περισσότερα υπάρχουν σε σχέση με την αντιμετώπιση της διαφθοράς από ότι σε άλλους τομείς. Έτσι λοιπόν όταν η σοφία της εντολής μου διατύπωσε τις αρμοδιότητές μου θέματα διαφθοράς δεν συμπεριλαμβανόντουσαν αλλά σίγουρα ισχύει αυτό ότι είναι εμπόδιο, είναι πρόσκομα για την επίτευξη όλων των στόχων που συζητήσαμε και αναφέραμε σήμερα το πρωί σε αυτή την ακρόαση. Δεύτερον, όσον αφορά την οικονομική κρίση, είναι πολύ δύσκολο να καλύψω τα θέματα με δύο λόγια. <clears throat> Βραχυπρόθεσμα είναι τρομερά τα πράγματα, μακροπρόθεσμα θα βελτιωθούν βραχυπρόθεσμα τρομερή κατάσταση, διότι όταν υπάρχει οικονομική κατάρρευση, οι ευάλωτοι οικονομικά πλήττονται σκληρότερα από όλους τους άλλους και ήδη ακούμε ιστορίες για την ε, ε, υποχρεωτική εργασία και πολλά άλλα πράγματα και στην συνολική αλυσίδα αυτών των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν πρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα όμως πιστεύω ότι η κρίση μάλλον θα έχει την ίδια επίπτωση όπως είχε η μεγάλη ύφεση ε, το κράχ ε, όσον αφορά την πολιτική αντιμετώπιση και προσέγγιση των θεμάτων στον βιομηχανοποιημένο κόσμο. Υπάρχει ε, μια αλληλουχία επιτακτική όσον αφορά την επανεξέταση του ε, συσχετισμού μεταξύ της αγοράς και των κρατών. Έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια. Πολλές από αυτές τις λεπτομέρειες από τεχνικά σώματα και οργανισμούς θα συζητηθούν για την ανάγκη αντιμετώπισης ρευστότητας, φερεγγιότητας, ε, εταιρική ε, ευθύνη ε, χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά εταιρικά θέματα. Δική μα δουλειά είναι να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε παρόντε σε όλα αυτά και δεν θα το αφήσουμε στου στενά επαείοντε ειδικού, α το πω έτσι, που δεν έχουν αυτέ τι συνιστώσει που έχουμε εμεί για τη δουλειά του. αλλά πάρα πολύ μεγάλη διαφορά μπορεί να επιτευχθεί στην αναθεώρηση των κανόνων και κανονισμών για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Όσον αφορά για παράδειγμα τι ευθύνε διευθυντών. Θα απαιτούσαμε από πλευρά των διευθυντών όσον αφορά τι υποχρεώσει του εναντί εταιρεία να λαμβάνουν υπόψη τι επιπτώσει ε, των δράσεων τη επιχείρηση στο περιβάλλον και τη κοινωνία. Βαθιέ διαφορέ σε σχέση με τη δυναμική των εταιριών και ε, ε, τι ευθύνε όσον αφορά τη λογοδοσία των διευθυντών. Αυτό ανοίγει μεγάλη δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, ευθύνης να υπάρχει διάρρηξη της ε, περαιτέρω της ε, υπόλοιπης δομής. Όλα αυτά μπορούν να έχουν τεράστια επίπτωση. Εκείνοι που κανονικά θα ε, συζητούσαν αυτά τα θέματα ως επαΐοντες δεν θα τα προσέγγιζαν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η δική μας φωνή και οι παρατήρησεις θα ακούγονται από πλευράς μας σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι η πιο αισιόδοξη συνιστόσα για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Θα υπάρξουν οι αλλαγές. Οι συζητήσεις αυτές, οι διαβουλεύσεις θα γίνουν και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θέματα αυτά κυρίως θέματα αηφορίας θα εισακουστούν. Και τέλος όσον αφορά το θέμα ποια είναι τα συμπεράσματα, τα μαθήματα που θα μπορούσαμε να συναγάγουμε από την εμπειρία της Γενέβης για παράδειγμα. Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί σύντομα αυτό το ερώτημα. Ένα ολόκληρο βιβλίο θα μπορούσα να γράψω και να το πουλήσω και να πάρω χρυσα... πολλά χρήματα. Όμως, σοβαρότερα τώρα, υπάρχουν, θα έλεγα, τρία στοιχεία που πιστεύω ότι μας διαφυλάτουν από, σε αυτή την διαδρομή ή σε αυτή την προσέγγιση. Ένα, η αιμονή στην εμπειρικότητα. Δεν ξεκινήσαμε με απαντήσεις έτοιμες, κομμένες και ραμμένες, αλλά με ερωτήσεις. Θέλαμε να μάθουμε και να γνωρίσουμε τι συνέβαινε, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, ποιες επιχειρήσεις, σε ποιες χώρες, ποιες προδιαγραφές εφαρμόζονται, ποιες άλλες δεν εφαρμόζονται, ποιες προσεγγίσεις είναι λειτουργικές, ποιες άλλες δεν είναι λειτουργικέ, ποιοι συνδυασμοί είναι καλύτεροι από άλλους. Είμαστε λοιπόν με ιδιαίτερη επιμονή και αιμονή εμπειρική στο χαρακτήρα μας. Ε, δοκιμάζαμε δηλαδή για να, να βρούμε τη σωστή προς, ε, απάντηση μέσω των σωστών ερωτήσεων. Και έτσι ένας ε, κοινός, ένας κοινός συνδυασμός στοιχείων ε, ετίθεντο επιτραπέζης που ήταν δεδομένα και δεν μπορούσε κανείς να τα αμφισβητήσει. Αυτό είναι η διάσταση των προβλημάτων. Αυτά τα πράγματα λειτουργούν, αλλά δεν λειτουργούν. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν την φύση τη ευρύτερη συζήτηση. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά εφ' εξή ε, στην ε, στενότερη έννοια τη διαφύλαξη ε, κάποιου συμφέροντο. Πρέπει μια κοινή βάση δεδομένων να λαμβάνεται υπόψη ω στοιχείο κίνηση. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, να στοχεύσουμε στοχοθετημένα σε ένα πλαίσιο <clears throat> για να υπάρξει ε, η διασφάλιση της ροής, της συνεκτικότητας και συνέχειας. Αυτό το πλαίσιο δεν είναι η απάντηση και λύση όλων των προβλημάτων, είναι μια κοινή βάση όμως που έχει δύο χαρακτηριστικά κύρια. Πρώτον, από όλους τους ε, εμπλεκόμενους τομείς ε, έχει ε, μια τροφοδοσία και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αφήνοντας πίσω την εταιρική κοινότητα διότι αυτονών η συμπεριφορά πρέπει να αλλάξει. Πρέπει λοιπόν η κοινότητα των επιχειρήσεων να συμμετάσχει. Πρέπει οι κυβερνήσεις να συμμετάσχουν και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αυτό που περιγράφουμε ως μια κοινή βάση, κοινά θεμέλια. Αυτά τα κοινά θεμέλια όμως και η κοινή βάση πρέπει να διαθρώνονται με, το, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκλείονται οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες. Όλοι να μπορούν να δουν τις προοπτικές μακροπρόθεσμα ανάλογα με τις πρόσθετες φιλοδοξίες ή ε, επιθυμίες τους ότι μπορούν να επιτευχθούν ξεκινώντας με, ως ε, κοινό θεμέλιο, ως κοινή βάση από αυτή την ε, αφετηρία ώστε να μην αποκλείονται προοπτικές και προ, άλλες εξελίξεις. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι σημαντικά. Η αιμονή στο να είμαστε ε, αποτελεσματικοί στην προσέγγιση με εμπειρικό χαρακτήρα δοκιμάζοντας να βρούμε το σωστό και δεύτερον να μην αποκλείσουμε ε, κινώντας από μια κοινή βάση τις θετικές προοπτικές στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο σας υποστηρίζει. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Η Μίκιο που είναι πολλές και δραστήριε Ελπίζουμε να συνεχίσουν να το κάνουν, παροτρύνοντας τους ε, μελλοντικού ευρωβουλευτέ για το θέμα αυτό. Μείνετε εδώ. Ήρθαν στο τέλο της συζήτηση δύο άτομα. Τους ξέρετε. Ο ένας είναι ένας γνωστός αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, κ. Μακμίλαν Σκότ, που συνοδεύεται από κάποιον που δεν γνωρίζετε, αλλά το οποίο το όνομα γνωρίζετε τον κύριο Έιμαν που τον παρακαλώ τον χειροκροτήσετε, έναν από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Αιγύπτιο, για τον οποίο το Κοινοβούλιο είχε δουλέψει πολύ για να απελευθερωθεί, απελευθερώθηκε το Φεβρουάριο. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι γι' αυτό και θέλουμε να τον καλέσουμε να πει δύο-τρεις φράσεις. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να πω ότι βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Λιγότερο από δύο μήνες ε, πριν από σήμερα είχα επιμείνει να μπορέσω να παρευρεθώ στην Ευρωβουλή ως το πρώτο βήμα αυτό εκτός Αιγύπτου στην, στην παρουσίασή μου και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσά σας ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήμουν φυλακισμένος ε, σε σχέση με την, ε, τα, τις προεδρικές εκλογές που είχαν γίνει στην χώρα μου Θέλω να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε για την ευκαιρία που είχα να σας συναντήσω και να μιλήσω μαζί σας στο Κάιρο και επενώ ιδιαίτερα την Ευρωβουλή για αυτό το ψήφισμα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το, συμβολικό χαρακτήρα του ψηφίσματος που είχε σημαντικότατη επιρροή και επίπτωση στην προσωπική μου περίπτωση και ζωή και στην περίπτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Όταν ήμουν φυλακισμένος διάβαζα τον Εμίρ Ζολά για τον Εμίρ Ζολά και τον ρόλο του στην υπόθεση Ντρέιφου ε, στην Γαλλία. Και τον υπερασπίστηκε τον Τρέιφους ο Ζολά. Διερωτήθηκα, υπάρχει κάποιος άλλος Εμίλιος Ζολά για μένα να με υπερασπιστεί εμένα ως κατηγορούμενο, ως κρατούμενο και είμαι υπερήφανος που μπορώ να πω σήμερα ότι βρήκα σε αυτό το υψηλό σώμα, εξέχον σώμα την Ευρωβουλή, εσάς πρόεδρε και τον αντιπρόεδρο επίσης κύριο Μακμίλαν Σκότ είδα σε εσά τον νέο Εμίλιο Ζολά συμβολικά. Νέους Εμιλίου Ζολά που βοηθούσαν εκείνους που υπέφεραν. Και νομίζω ότι η θέση αυτή είναι ακριβώς ε, η ευθύνη που έχω να το εκφράσω αυτό και για το ότι κατάφερα να αποκτήσω μέρος της ελευθερίας μου. Δεν απέκτησα όμως και δεν ανέκτησα όλα μου τα δικαιώματα ακόμα. Μέρος της ελευθερίας μου όπως είπα ανέκτησα Υπάρχουν όμως εκατοντάδες και χιλιάδες, ε, μυριάδες στον αραβικό κόσμο που είναι θύματα, αθώα θύματα δεσποτείας και αυταρχικών καθεστώτων. Έχω καταλόγους ονομάτων στη Συρία, στη Δαμασκό, στην Αίγυπτο. Είναι όλοι αυτοί θύματα στρατιωτικών δικαστηρίων. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη εκεί ε, και δύο οι οποία ήταν bloggers ε, και μάλιστα σε σχέση με την δραστηριοποίησή τους ε, τυπώνοντας και ένα βιβλίο προσάχθηκαν στα δικαστήρια και καταδικάστηκαν. Υπάρχουν άλλοι bloggers όπως ο Καρίν Άνερ που ήταν από το κόμμα μου που αποκλείστηκε, εκδιώχθηκε από το Πανεπιστήμιο και βρίσκεται ακόμα στη φυλακή επειδή συνέταξε τις, τις απόψεις του και δημοσιοποίησε εξ ονόματος των διοκόμενων. Επίσης ο Ιμπραχήμ ο οποίος ε, διώκεται ακόμα και δεν μπορεί να επιστρέψει στην ε, ε, Αιγυπτό Ανβάρ Ιμπραχήμ για όλους αυτούς και εξ ονόματος τους θα ήθελα να σας πω ότι συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα είναι εκείνη η οποία θα κάνει το καθήκον τη απέναντι σε αυτούς και σε εμάς διότι η Ευρώπη είναι η πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλά περιμένουμε και προσδοκούμε από εσάς όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας, γενικότερα. Και πάλι σας ευχαριστώ βαθιά κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ βαθιά για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας προσφωνήσω απευθύνοντάς σας αυτές τις παρατηρήσεις μου, αυτά τα λόγια και να παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας και ελπίζω ότι πάντα θα είμαστε υπέρ τη ελευθερία όλων των θυμάτων παντού για όλους τους κρατούμενους συνείδησης ε, διαφωνούντες παντού, όχι μόνο στην Αίγυπτο και στον Αραβικό κόσμο. Σας ευχαριστώ και... Ευχαριστώ κύριε Μαϊνού. Θα προσπαθήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρήσουμε και να σεβαστούμε τις προσδοκίες ατόμων όπως εσείς που ζείτε σε δύσκολες χώρες προς τιμήν των προσκεκριμένων μας. Σας καλώ σε ένα ποτηράκι